Dear colleagues, I would like to start the meeting because we have a lot of points actually for this afternoon. I would like to start with. Θα γίνει τώρα η παρουσίαση της ΙΤΑ συνεδρίασης. Έχουμε τον κύριο Κόρκα που είναι ο επικεφαλής του σχετικού τμήματος και την κυρία διοικητική υπάλληλο από, την διοικητή, από τη Γενική Διεύθυνση ITEC. Για αυτή την υπηρεσία που θα μας επιτρέπει να έχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερα, αν όχι όλα, τα ένιγραφα των συνεδριάσεων. Ορίστε λοιπόν σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνεται να σας παρουσιάσουμε το ΙΤΑ συνεδρίαση. Το ΙΤΑ συνεδρίαση είναι ένα εσωτερικό εργαλείο που πολλοί από εσά το ξέρετε ήδη γιατί το δοκιμάσαμε και στην προηγούμενη θητεία. Τώρα όμως είναι σε χρήση σε ολόκληρο το κοινοβούλιο και διατίθεται σε, για όλο το προσωπικό και τους ε, ευρωβουλευτάς. Είναι εφαρμογή που δίνει σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα των συνεδριάσεων σε όλα τα μηχανήματα. Smartphone, κινητό υπολογιστή, αλλά το καλύτερο μηχάνημα είναι το iPad. Μάλλον ήδη ξέρετε ότι τα μέλη θα λάβουν τα iPads των τους επόμενους μήνες και τότε θα μπορείτε όλοι να τα χρησιμοποιείτε πιο εύκολα από ό,τι τώρα. Λοιπόν, η ήττα συνεδρίαση είναι, ε, επιτρέπει γενικά να επωφελούνται όσοι κινούνται πολύ και χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάνε τους χαρτοφύλακες με τα χαρτιά τους. Βεβαίως και τα χαρτιά και τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν το καθένα τα υπέρ και τα κατά τους. Βλέπ, θα σας πω ποια είναι τα υπέρ του e-meeting όταν θα το δείξουν οι διαφάνειες ο συνάδελφος εδώ. Είναι μέσα στα πλαίσια του intranet το AFCONET η τα συνεδρίαση για την Επιτροπή σας ειδικά Θα σας κάνουμε μία επίδειξη και μετά έχουμε εδώ τον γρήγορο αυτό οδηγό που έχετε μπροστά στα έδρανά σας για να δείτε τις οδηγίες και μετά. Αν έχετε το iPad σας να το ανοίξετε και να παρακολουθήσετε την επίδειξη για να δείτε και μόνοι σας πώς δουλεύει. Μετά την επίδειξη θα απαντήσουμε οτιδήποτε απορίες μπορεί να τεθούν και φυσικά και για πιο και ιδιαίτερος άμα χρειαστεί. Με την ε, άδεια της Προέδρου δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου με τις διαφάνειες. Ευχαριστώ πολύ. Η εφαρμογή λοιπόν αυτή είναι εφαρμογή διαδικτύου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να εγκαταστήσετε τίποτα για να έχετε πρόσβαση. Με αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Να, θα σας το γράψω εδώ και μπορείτε και εσείς να το γράψετε πάνω στα μηχανήματά σας. Εγώ το επιδεικνύω σε iPad αλλά δουλεύει και σε άλλα μηχανήματα. Η εφαρμογή είναι εσωτερική και πρόσβαση έχουν μόνο οι βουλευτές και το προσωπικό και οι βοηθοί. Θα δώσω το δικό μου όνομα χρήστη, όχι το κανονικό βέβαια. Χρησιμοποιήστε και εσείς το δικό σας και το σύνθημα. Την πρώτη φορά που μπαίνετε στην εφαρμογή βλέπετε αυτή την οθόνη. Είναι βοηθάει, πατήστε το Start Τώρα είμαι μέσα στην εφαρμογή. Βλέπετε ότι είναι εσωτερική εφαρμογή. Πάνω αριστερά έχετε την επιλογή των γαλωσσών. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Κοντά εκεί είναι οι επιτροπές και ισχύει για όλες τις επιτροπές. Ας πούμε εδώ αύκο. Το σύστημα παίρνει τις τελευταίες εκδοχές των εγγράφων που αφορούν την κάθε συνεδρίαση και μπορώ να τα δω και, δω και προηγουμένων συνεδριάσεων μέχρι το 2010. Όλη η πληροφόρηση αυτή παραμένει εσωτερική και πριν τη συνεδρίαση και μετά και στους διαδρόμους και στο δρόμο. Εδώ δεξιά έχετε την ημερήσια διάταξη και όταν έχει ένα συν στα θέματα και πατήσετε το συν έχετε περαιτέρω πληροφορίες, ονόματα, έγγραφα. Πάνω δεξιά έχουμε την άποψη, την όψη μόνο των εγγράφων Μπορεί κανείς κάποτε σε κάποια συνεδρίαση να θέλει να ε, δώσει, να στείλει αυτό το έγγραφο και σε άλλον. Γίνεται από αυτό το, αυτή την επιλογή 5. Και αν θέλετε τίποτε προσθήκες υπάρχει ένα έγγραφο που το επιτρέπει. Τώρα πάλι στην μερίσια διάταξη θα σας δείξω τι μπορεί να γίνει. πούμε ότι πάμε στο σημείο 7, έγγραφα εργασίας, πάλι για όλες, σε όλες τις γλώσσες, ας πούμε εδώ Ιταλικά. Το σύστημα ανοίγει την τελευταία εκδοχή, αυτή είναι η τελευταία εκδοχή, μπορώ να το διαβάσω. Τώρα φανταστείτε ότι θέλετε να κάνετε σημειώσεις. Τότε χρειάζεται να βοηθηθούμε από μια εξωτερική εφαρμογή κάποια. Εδώ έχω την δωρεάν εφαρμογή που υπάρχει και από την οποία μπορώ να σημειώσω πράγματα στο έγγραφο που διαβάζω. Να υπογραμμίσω, να σβήσω και να γράψω σχόλια. Λοιπόν, όταν είμαι ικανοποιημένο από τις αλλαγές, μπορώ να τις στείλω σε συναδέλφους, τους βοηθούς και όλα όσα πρόσθεσα στο εγγραφό μου θα σωθούν με μορφή PDF και μπορώ να τα στείλω σε όποιο θέλω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σενάριο της χρήσης του ΙΤΑ συνεδρίαση. Να διαβάσω, να αλλάξω, να στείλω. Επίσης θέλουμε να σας δείξουμε ότι για κάθε επιτροπή έχουμε το e-committee Site δηλαδή σε ένα μέρος όλα τα έγγραφα που αφορούν τη δουλειά μιας επιτροπής είναι άλλη σελίδα την οποία οργανώνει κάθε επιτροπή και έχει πληροφορίες για τη δουλειά της Επιτροπής. Εδώ ας πούμε έχουμε πληροφορίες για τα μέλη, το Προεδρείο, τους βοηθούς. Εδώ τώρα σας φαίνεται ίσως αργό γιατί γίνεται με το wifi αλλά σε υπολογιστή κανονικό πάει πολύ γρήγορα λοιπόν. Εδώ αριστερά έχουμε ένα κεφάλαιο που λέγεται Work in Progress και δίνει πληροφορίες για τις τρέχουσες εκθέσεις. Α, δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω. Δεν βλέπω κανένα έγγραφο εδώ. αλλά ας πούμε ότι πάω σε άλλη επιτροπή για να δω σε άλλη να δω αν πάω σε αυτή την συνεδρίαση μπορώ να δω και την ημερήσια της διάταξη και εδώ πάλι μπορώ να την εξαγάγω ως γεγονός στο ημερολόγιο ή όπως έκανα πριν στο e-meeting να δω την ε, ημερήσια διάταξη. Υπάρχει λοιπόν το e-meeting, υπάρχει και το e-committee. Εδώ είναι το ίδιο στυλ. Αν χρησιμοποιήσω μια άλλη επιτροπή, την NOM ας πούμε, η ίδια οργάνωση, έχουμε τις πληροφορίες και αν θέλω να πάω στη νομική με το e-committee πάλι το ίδιο στυλ είναι. Παρουσιάζουμε με τον ίδιο τρόπο τις πληροφορίες για να μην ξενίζεται ή ξυπάζεται ο χρήστης. Εδώ ας πούμε στο work in progress, στα σχέδια εγγράφων, μπορώ να δω όλες τις εκθέσεις ή σχέδια εκθέσεων της νομικής, τις γνωμοδοτήσεις, τις ψηφοφορίες, τον διοικητικό υπάλληλο, τους κοιόδης. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι η παρουσίαση των δύο ψηφοφοριε τον ή εφαρμογών σκιωδης επιτροπή και ή τα συνεδρίαση. Και αν έχετε σχόλια παρακαλώ να μας τα κάνετε. Ε, δεν έχουμε όμως χρόνο για ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και η υπηρεσία βοηθητική αν κανείς θέλει να σας πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει. Μάλιστα, μάλιστα, όλα εδώ είναι. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει ποτέ να καταργηθεί πλήρως το χαρτί και θα είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό σύστημα. Όχι, ο καθένας θα αποφασίσει μόνος του αν θέλει τα χαρτιά ή όχι. Θα συνεχίσουν τα χαρτιά δηλαδή. Μάλιστα. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει καμιά απόφαση κατάργησης του χαρτιού. Άρα ο καθένας θα αποφασίσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κατάλαβα ότι είστε διαθέσιμοι αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιάς μας διάταξης που είναι η πληροφόρηση για τα αυτά που αποφασίσαμε στους συντονιστάς. Επιβεβαιώσαμε τις εκθέσεις που πρότειναν οι πράσινοι για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία εισηγητής Ντουράν επίσης αποφασίσαμε για την κατανομή των γνωμοδοτήσεων ε, από άλλες επιτροπές, προς άλλες επιτροπές την ετήσια έκθεση 12 για την επικουρικότητα πήγε στους συντηρητικούς. Η 30 και 31η έκθεση για την επιτήρηση του κοινωτικού δικαίου του FDD. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στους σοσιαλιστάς και για το ΕΛΚ οι συστάσεις της Κομισιόν για το TTIP. Επίσης αποφασίσαμε ότι τα αιτήματα αλλαγών του κανονισμού που προέρχονται από δύο βουλευτές, De Jong και Γκέρενς, δόθηκαν στην ομάδα εργασίας που θα μας κάνει συστάσεις δεχτήκαμε τις ημερομηνίες των ακροάσεων για τα μαθήματα από την εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών 26 Φεβρουαρίου. Ε, θεσμικά και ευτυχές για τη διακυβέρνηση 31 δηλαδή Μαρτίου για το μέλλον της Ένωσης 16 ε, Απριλίου και τις ημερομηνίες για τα λεγόμενες μήνυα ακροάσεις μέσα στα πλαίσια κανονικών συνεδριάσεων χωρίς να πληρώνονται οι εμπειρογνώμονες πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απόφαση του δικαστηρίου το Δεκέμβριο και μετά για την πρόσβαση της Ένωσης Χάρτα των Θεμελιο... Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον Ιούνιο μετά πληροφόρησα τους συντονιστάς και σας πληροφορώ και σας ότι είναι πολύ πιθανό να γιοργανωθεί κοινή ακρόαση με τη νομική και τη δημοσιονομική μαζί μας για την λογοδοσία αλλά η απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί επίσημα. Επίσης η ζήτησε να έχει το δικαίωμα να ορίσει focal point για την ισότητα των φίλων για την ΑΦΚΟ και ο κύριος Γεώργιος Κατρούγκαλος θα είναι ο εκπρόσωπος της ΑΦΚΟ για αυτό το θέμα. Να, αυτά αποφασίσαμε στους συντονιστάς. Τώρα το σημείο 7 της σημερινής διάταξης, ο Ριχάρτος Κόρμπετ θα το χειριστεί. Είχαμε αποφασίσει να ορίσουμε εισηγητή για τις ακροάσεις και τις μεταακροάσεις τον Ρίτσαρντ Κόρμπετ τον Ιούλιο και τώρα έχουμε το έγγραφο εργασίας του για τις ακροάσεις του 14 και με βάση αυτό το έγγραφο εργασίας θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να γράψουμε και έκθεση ιδίας πρατοβουλίας. Σήμερα θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το έγγραφο εργασίας του Ριχάρδου, ο οποίος έχει και το λόγο και λέγεται Κόρμπετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το έχουν λάβει οι συνάδελφοι μέσω αυτού του υπέροχου ηλεκτρονικού συστήματος αλλά και σε έντυπη μορφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έγγραφο εργασία για κάποιες πρώτες ιδέες ε, για να λύσουμε κάποιες ιδέες για να το βελτιώσουμε την επόμενη φορά. Τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, πού πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες μας. Μετά από το έγγραφο μετά θα περάσουμε σε ένα σχέδιο έκθεσης. Η έκθεση αυτή, αν εγκριθεί, θα ε, καταλήξει στα συμπεράσματά μας που ίσως σε κάποιες περιπτώσεις απαιτήσουν συζητήσεις με άλλα θεσμικά όργανα ή ίσως σε κάποιες περιπτώσεις απαιτήσει αλλαγές του κανονισμού οπότε μετά θα πρέπει να τα δει ομάδα κανονισμού και σε άλλες περιπτώσεις ίσως απλά καταλήξει σε κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Θα το δούμε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την εμπειρία μας. Τα έγγραφα βεβαίω υπενθυμίζουν πρώτα απ' όλα το υπόβαθρο της υπόθεσης είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα από τη συνθήκη χωρίς να ζητήσουμε κανονισμό ή διακυβερνητική οι κυβερνήσεις είπαν πως το Κοινοβούλιο είπε πριν ψηφίσει επί της Κομισιόν να έρχονται οι επιτροπές, η επίτροποι εδώ πέρα υποψήφοι για μια τρίωρη δημόσια κουράση. Το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια. Είναι κάτι το εδρεωμένο, κανείς δεν το αμφισβητεί πλέον, κάτι το οποίο συνέβαινε στην αρχή, αλλά δεν συμβαίνει πλέον. Και αυτό γενικά θεωρείται κάτι το θετικό. Δηλαδή ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με κανέναν υποψήφιο επίτροπο, καλό θα ήταν και πάλι από πλευράς διαφάνειας να γνωριστούμε με τους μέλους επιτρόπους, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές τους και βεβαίω πάντα υπάρχουν κάποια προβλήματα και, και αυτή τη φορά και την προηγούμενη υπάρχει πάντα μια αλλαγή στη σύνθεση της Κομισιόν όπου κάποιος, κάποια υποψήφιος ε, δεν άρεσε στους συναδέλφους. Αλλά πέρα από αυτό σημαίνουν και άλλα υποσχέσεις, ε, δεσμεύσεις. Ε. Δεσμεύονται οι επίτροποι για κάποια πράγματα, γίνονται διευκρινήσεις, αλλαγές χαρτοφυλακίων, οπότε πάντα κάτι το θετικό υπάρχει, αλλά πάντα ε, μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Τα έγγραφά μου Εάν δείτε τη σύνοψη εδώ πέρα, τα στατιστικά στοιχεία κτλ. Θα δείτε το σημείο 7 που λέγεται ζητήματα. Και έχω προτείνει εγώ 7 πράγματα για να ξεκινήσει η συζήτηση, ε, σημεία στα οποία θεωρώ πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτά απλά λοιπόν για να ξεκινήσει η συζήτηση. Το πρώτο θέμα αφορούσε τον χρόνο. Ε, είχαμε πιεστεί κάπως αυτή την ε, φορά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί από τώρα τα κράτη-μέλη απλά όρισαν αργά τους επιτρόπους. Μπορούμε να το συζητήσουμε θα μπει μια προθεσμία να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν νωρίτερα προτάσεις. για να μας θέλουν κάποιοι. Γιατί βεβαίως ε, αν είχαμε μια προθεσμία θα έπρεπε και να την τηρήσουν. Το δεύτερο θέμα είναι εσωτερικό. Μία ακρόαση έγινε από τη διάσκεψη των Προέδρων. Όμως ο κανονισμός λέει πως οι επιτροπές κάνουν τις ακροάσεις. Οπότε δεν έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό αυτή η ακρόαση. Έτσι, αν το δούμε ε, αυστηρά. Βεβαίως υπήρχε σοβαρός λόγος, πρόκειτο για την ε, ακρόαση του κυρίου Τίμερμανς, ο οποίος είχε πολλές οριζόντιες αρμοδιότητες ως πρώτος αντιπρόεδρος. Οπότε εντάξει δεν ξέρω τι θα γινόταν, θα ήταν με 4-5 επιτροπές. Ήταν λογικό να γίνει στην διάσκεψη των Προέδρων ε, παρουσία όλων των μελών, έτσι, όλων των βουλευτών. Αλλά πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Θέλουμε να γίνεται μονίμως αυτό το πράγμα ε, ή μπορούμε να πούμε όχι λάθος ήταν αυτό και πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία. Οπωσδήποτε στο μέλλον εάν ε, αντιμετωπίσουμε κάποια διαρθρωτικά ζητήματα και έχουμε αντιπρόεδρο με οριζόντιες αρμοδιότητες θα πρέπει ίσως να δούμε αυτή την επιλογή. Το τρίτο ε, ζήτημα και το, ένα από τα σημαντικότερα κατά την άποψή μου αφορά το ύφο των ερωτήσεων. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε πως κάθε ακρόαση θα έχει 45 ερωτήσεις του ενός λεπτού ε, και μετά απαντήσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως αυτό είναι λάθος. Λιγότερες ερωτήσεις χρειάζονται, αλλά με δυνατότητα ε, και άλλων ερωτήσεων. Να υπάρχει έτσι μια συζήτηση. Εξάλλου στόχος δεν είναι να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές. Ο στόχος ε, είναι να υπάρξει ακρόαση και να υπάρξουν ερωτήσεις ε, προς ε, τον Επίτροπο και να υπάρχει δυνατότητα για επερώτηση αμέσως αφού δοθεί η αρχική απάντηση. Βεβαίως, αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι άποψη που συμμερίζονται αρκετοί. Τέταρτο ερώτημα, σημείο 7D στο έγγραφο εργασία είναι το θέμα της αξιολόγησης. Θα πρέπει να υπάρχει και λίγος χρόνος για τις ομάδες να κάνουν μια συζήτηση ε, για τα θέματα αυτά Τα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν στη διάρκεια της αξιολόγησης των συνεδριάσεων είναι τι θα γίνει αν δεν συμφωνούν οι συντονιστές ομόφωνα. Διότι οι κανόνες λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση για το κατά πόσον είναι κατάλληλος ή όχι ένας υποψήφιος. Κάποιες φορές ε, σχεδόν όλες οι ομάδες πίστευαν ότι όντως αυτό συνέβαινε, αλλά υπήρχαν μία-δύο πολιτικές ομάδες που διαφωνούσαν και βρέθηκαν κάποιες ευέλικτε ε, ε, λύσεις, για παράδειγμα να γραφεί μία επιστολή που να λέει ότι υπάρχει συνένεση, αλλά διαφωνεί τάδε η δίνα πολιτική ομάδα ότι ο τάδε ε, υποψήφιος είναι αποδεκτή ή όχι. Ε, αυτή είναι ερμηνεία των κανόνων, δεν είναι κατά γράμμα ε, εφαρμογή αλλά σε κάποιε περιπτώσεις έπρεπε να ρωτήσουμε κάποιε περισσότερες ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσεις και σε μια περίπτωση ε, κλήθηκε και πάλι ο Επίτροπος για δεύτερη ακρόαση, παρά το γεγονός η, ότι οι κανόνες αναφέρονται σε μία ακρόαση. Βέβαια, ε, επισήμως την αποκαλέσαμε μια δεύτερη συνεδρίαση, αλλά στην ουσία όλοι την αποκαλούν δεύτερη ακρόαση. Εγώ προτείνω να βάλουμε μια τάξη και ε, πρότεινα εκεί τι θα μπορούσε να συμβεί. Αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση ή ομόφωνη απόρριψη, ε, να μπορέσουμε να έχουμε μία επιστολή και να ε, τα γράψουμε αυτά και τέρμα υπόθεση. Και προτείνω μια ιεράρχηση. Αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, τότε θα πρέπει να το λέει η επιστολή. Αν είναι ισομερή η κατανομή ή αν υπάρχει κάποια ο επίμαχο ζήτημα, τότε θα μπορούσαν να υπάρχουν δυνατότητα για επιπλέον επιλογέ. Είτε περαιτέρω ερωτήσει, δεύτερον μια δεύτερη ακρόαση, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι εξαιρετική περίσταση, μόνο με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Και τέλο, ω τελευταία λύση, τότε περνάμε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή. Και γιατί λέω ψηφοφορία ότι θα πρέπει να είναι η ίστατη λύση διότι, όπως γνωρίζουμε, επισήμως βάσει της συνθήκης, το Κοινοβούλιο στο σύνολό του ψηφίζει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο σύνολό της. Ναι. Οι ψηφοφορίες για τον κάθε επίτροπο και ψηφοφορίες σε κάθε επιτροπή για κάθε επίτροπο δεν έχουν καμία νομική ε, υπόσταση. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αν περάσουμε σε αυτή την εναλλακτική λύση, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Επομένως, δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι το οποίο θα είναι δεδομένο και θα είναι συνήθεια μετά από κάθε ακρόαση, κάθε επιτρόπου να γίνεται ψηφοφορία στην Επιτροπή. Γι' αυτό ακριβώς και πρότεινα να υπάρχει μεν αυτό το ενδεχόμενο, αλλά να είναι σαφώς η ίστατη λύση όταν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και βεβαίως, επειδή δεν θα συμβαίνει κάθε φορά, θα έχει και την αντίστοιχη πολιτική βαρύτητα, την πολιτική βαρύτητα που του αναλογεί. Πέμπτο θέμα, πολύ απλό. Οι κανόνες μας αυτή τη στιγμή λένε ότι θα πρέπει να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 24 ώρες μετά την ακρόαση αλλά ορισμένε φορέ οι αξιολογήσει καθυστερούν πολύ περισσότερο. Επομένω δεν μπορεί να γίνει. Επομένω άλλαξα τον κανόνα και έλεγα λογικά θα πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρε μετά την αξιολόγηση. Δηλαδή γίνεται η αξιολόγηση, άρα πρέπει να δημοσιευθεί ε, εντό 24 ώρου. Το έκτο θέμα το αποκαλώ οριζόντια θέματα και αυτό γιατί στις ακροάσεις κάποιες φορές τίθενται ερωτήσεις που πραγματικά δεν μπορεί να απαντήσει ο υποψήφιο, γιατί είναι μια ερώτηση που αφορά το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτήσει του τύπου. Ε, ποια είναι η σχέση μεταξύ αντιπροέδρων και ε, των υπολείπων επιτρόπων, που είναι μια ερώτηση που ανέκυψε αρκετέ φορέ. Ερωτήσει που έχουν να κάνουν με την ισορροπία όσον αφορά άνδρε-γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υποψήφιο επίτροπο δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτέ τι ερωτήσει. Αυτέ είναι ερωτήσει που μόνο ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να απαντήσει. Αλλά ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακρόαση γιατί τον έχουμε κλέξει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, προβλέπεται και μια συνεδρίαση στη διάσκεψη των Προέδρων, ίσως ε, ανοιχτή επιτροπή με τον ε, εκλεγμένο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στα θέματα τα οποία δεν θα μπορεί να απαντήσει ο κάθε Επίτροπος ξεχωριστά. Έβδομη παρατήρηση. δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Ιδιαίτερα με κάποιον επίτροπο, ένα συγκεκριμένο, η δήλωση των οικονομικών συμφερόντων του δεν ήταν η κατάλληλη, δεν mm. συζητήθηκε καταλήλων. Αυτό πάντα παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί τη ουσία για το θέμα αυτό, και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξετάζει κατά πόσον η δήλωση οικονομικών συμφερόντων που έκανε ο επίτροπο συνάδει με του κείμενους κανόνε και διατάξει επί του θέματο. Mm. Δεν μπόρεσαν να πάνε πέρα από αυτό. Πολλά μέλη θεώρησαν ότι θα έπρεπε να, να πάνε πέρα από αυτό, διότι αυτή ε, είναι μια υπόθεση η οποία υποτίθεται ότι ε, ε, ενήχε και μεταφορά μετοχών σε μέλη της οικογένειας του εν λόγω επιτρόπου. Για να μπορέσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε καταλήλως το θέμα, πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για το τι πρέπει να δηλώνουν οι επίτροποι στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Και αυτό απαιτεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει βέβαια ε, ολόκληρη επιχειρηματολογία υπέρ ε, και υπάρχουν και επιχειρηματολογία βεβαίω κατά, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί μόνο μερό. Θα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υπάρχει έκθεση εν ευθέτω χρόνο στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει και η Επιτροπή μα, δεν είμαι βέβαιο, και θα πρέπει να υπάρχει διεύρυνση του τι θα πρέπει να περιλαμβάνει δέρο οικονομικών συμφερόντων στο μέλλον προσωπικώ φρονώ ότι αν το ζητήσουμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λογικά θα πρέπει να το ζητήσουμε και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης και για τις δικές μας δηλώσεις. Mm. Και τα μέλη θα πρέπει να το γνωρίζουν ότι αν επιμείνουμε και θέλουμε οι Επίτροπη να ε, περιλαμβάνουν περισσότερα πράγματα στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, λογικά, για λόγους διαφάνειας και δικαιοσύνης και ισότητας, να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες και για μας, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις δικές μας δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων. Και αυτό πρέπει να το περιλαμβάνει και ο δικός μας ο κανονισμός. Ε, αυτό νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι θέματα τα οποία ε, ενετόπισα και θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ε, θα σκεφτούν ίσως οι συνάδελφοι. Αφού το έγραψα την έκθεση μου το επεσήμανε και κάποιος, υπάρχει ένα σημείο ε, προθεσμία για ε, τροπολογία γιών των κρατών μελών είναι δυνατόν να ζητάμε από κάθε κυβέρνηση να ορίζει δύο υποψηφίους επιτρόπους, έναν άνδρα και μία γυναίκα και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος τη Επιτροπής να αποφασίζει. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε, είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο κειμένου μου, αλλά ίσως θα έπρεπε να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ρίτσαρντ. Πριν ε, ξαναδώ στο λόγο να σας πω πως οι συντονιστές ακόμα δεν έχουν ε, λάβει απόφαση, αλλά προς τα εκεί πάμε. Αντί δηλαδή να πάμε σε αναθεώρηση του κανονισμού, καλό είναι να γίνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για να ακούσουμε και τα σχόλια της Γιούρη. Ε, για να συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές να έχουμε και αυτή την πτυχή. Ελπίζω λοιπόν να ληφθεί αυτή η απόφαση σύντομα. Εν τω μεταξύ ο κύριος Πρέντα από ό,τι κατάλαβα. Έχει κάποιες απόψεις που θα ήθελε να εκφράσει έτσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας εκεί με τα γυαλιά για την παρουσίασή του θα κάνω και εγώ μερικά γενικά σχόλια για να συνεχίσει η συζήτηση έτσι. Πρόκειται βέβαια για πολύ πλούσιο κείμενο με πολύ βαθιά ανάλυση της διαδικασίας των ακροάσεων και η προσέγγιση του το καθιστά ένα αξιοσημείωτο εργαλείο για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για το θέμα των ακροάσεων των επιτηρόπων. Τώρα για τη βελτίωση των διαδικασιών έχει ενδιαφέρουσες προτάσεις επίσης. Και θα σχολιάσω σύντομα αυτά τα θέματα. Για το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων, πρώτο θέμα, πρέπει πράγματι να έχουμε μια ημερομηνία εκ των προτέρων ώστε να μπορούν τα κράτη να γνωστοποιήσουν και αυτά εν καιρό τον υποψήφιο. Και μετά θα θυμάστε ότι φέτος το Βέλγιο είχε αποφασίσει την προηγουμένη μόλις της ακρόασης το όνομα του υποψηφίου και έπρεπε να διαλέξουν άντρα ή γυναίκα. Εάν η βελγική κυβέρνηση δεν όριζε γυναίκα, τότε η Κομισιόν στο σύνολό της θα αντιμετώπιζε δυσκολίες γιατί ο Γιούνκερ είχε αποφασίσει ότι θα είχε 9 γυναίκες η Κομισιόν για τις κυβερνήσεις που έκαναν δύο προτάσεις όπως και εγώ όπως και η δική μου χώρα η Ρουμανία, ο Γιούνκερ διάλεξε την σοσιαλίστρια και όχι τον χριστιανοδημοκράτη για να φτάσει την ποσόστοσή του για τις γυναίκες. Επομένως εδώ είναι η χρησιμότητα της διορίας. Οι Βέλγοι δεν σεβάστηκαν την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί και δεν φτάνει Βέλγοι βέβαια μόνο, όρισαν τον Επίτροπο μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς τους. Ήταν τυχαίο. Γενικά όμως βρίσκω ότι αν συμφωνήσουμε ότι θα γίνονται οι εκλογές τέλη Μαρτίου και όχι αρχές Ιουνίου, ώστε να μπορούμε στο δυνατόν συντομότερα να συμφωνήσουμε και για την Κομισιόν, τότε θα μπορούσα να κάνω μια προσπαθιούλα και τα κράτη-μέλη για να σεβαστούν μια διορία χωρίς να τα βλέπουν όλα εθνικά. Επαναλαμβάνω, οι Βέλγοι όρισαν τον επίτροπό τους μέσα στα πλαίσια της γενικότερης διαπραγμάτευσης για την κυβέρνηση που έγινε, γιατί οι εκλογές γίνονταν την ίδια μέρα με τις εθνικές. Δεύτερον, συμφωνώ ότι η ακρόαση του Τίμερμανς αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή και σε παραβίαση των διαδικαστικών κανόνων. Ε, όλοι μας μας αρέσει ο Τίμερμανς, αλλά ήταν αυτοσχεδιασμός αλλά αυτά. Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με όλη τη δουλειά των υπολείπων επιτροπών. Τέτοια προσπάθεια για να γίνουν πολύ αυστηρές και ακριβείς ακροάσεις, ενώ στην περίπτωση του Τίμερμαν σε πρόκειτο για αυτοσχεδιασμούς. για την αποτίμηση των υποψηφίων, σημείο Δέλτα, συμφωνώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες, να βασιστούμε δηλαδή στο ότι μπορεί να πάνε τα πράγματα και πολύ άσχημα δηλαδή να υπάρξει καταστροφή και όχι να βασιστούμε στην καλύτερη δυνατή υπόθεση. Και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρξει μια, ένας καλύτερος συνδυασμός των επιστολών από τις διάφορες επιτροπές. Κατά τα υπόλοιπα, για το γάμα, το ύφος των ερωτήσεων, ο εισηγητής λέει να μειωθούν 40, από 45 σε 25 οι ερωτήσεις και να είναι ερώτηση και απάντηση συνεχώς. Και το δικαιολογεί αυτό λέγοντας ότι ο στόχος δεν είναι να εκφραστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για να προετοιμαστούν καλύτερα οι ακροάσεις με συντονισμό λέει μεταξύ των ομάδων και για τις ερωτήσεις. Εδώ έχω δύο αντιρρήσεις. Είμαι και εγώ συντονιστής στην ΕΠΕΞ και οι συνάδελφοί μας εκεί απογοητεύτηκαν γιατί δεν είχαν χρόνο ομιλία στις ακροάσεις για τον Κερίνη και τον Χάν. Και επομένως η δική μας λύση ήταν να χωρίσουμε σε δύο ίσες ομάδες, σχεδόν ίσες, 21 μέλη του ΕΛΚ και δεν χωρίζονταν ακριβώς τα δύο, 11 και 10 στις δύο ακροάσεις, αλλά ως συντονιστής εγώ μπόρεσα να μιλήσω και στις δύο ακροάσεις, οι άλλοι όμως αναγκάστηκαν να επιλέξουν. Και δεν είναι εύκολο γιατί οι βουλευτές θέλουν να εκφραστούν ανάλογα με τις ικανότητές των. Διότι οι βουλευτές θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή της θητείας τους οι ακροάσεις, δεν είναι κάτι δευτερεύον. Όταν έρχονται λοιπόν για ακρόαση θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό και όχι μία συνάντηση σαν τις άλλες. Να το προσέξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται συγκέντρωση της προσοχής στα ουσιώδη, αλλά ταυτόχρονα οι βουλευτές πρέπει να μπορούν να ασκήσουν αυτό το σημαντικό τους δικαίωμα. Να μην δώσουμε περισσότερη σημασία στους επιτρόπους από τους συναδέλφους μας. Πρώτα στους συναδέλφους και στο πώς βλέπουν την ακρόαση. Επίτα δεν συμφωνώ ότι πρέπει εκ των προτέρων να συνεννοούνται οι ομάδες. Καλά για αριθμούς, για ονόματα κτλ, για τη σειρά, Εντάξει, αλλά για το περιεχόμενο όχι, γιατί είναι πολιτικές οι ακροάσεις, πολιτικές. Η ύπαρξη του μεγάλου συνασπισμού άλλαξε πολύ το χαρακτήρα των ακροάσεων. Είμαι λοιπόν κατά της ιδέας μια συνεννόησης ενός συντονισμού επί της ουσίας, γιατί είναι πολιτικές οι ακροάσεις και πρέπει να παραμείνουν αντιπαράθεση. Τώρα για το F. Οριζόντια θέματα εξορρόπηση των φίλων κλπ. Ο εισηγητής μας δίνει μερικές ιδέες και θα ήθελε η συνάντηση του Προέδρου της Κομισιόν με τη διάσκεψη των Προέδρων να γίνεται στο τέλος των ακροάσεων πριν, πριν, εγώ νομίζω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και ένα άλλο οριζόντιο θέμα, η ανταπόκριση μεταξύ της εσωτερικής μας δομής και της δομής της Κομισιόν. Η ιδέα του Γιούνκερ να εξορθολογιστεί η δουλειά της Κομισιόν είναι σωστή, αλλά δημιούργησε πολλούς πανακεφάλους. Οι ακροάσεις με τρεις-τέσσερις επιτροπές μαζί δεν είναι εύκολες. Είναι δύσκολο να τις διαχειριστούμε και αν κάνουμε αυτό που λέτε με 35 ερωτήσεις φανταστείτε πού μπορεί να φτάσουμε ε, 25 μάλλον ερωτήσεις τέσσερις επιτροπές με 25 ερωτήσεις θα γίνει πόλεμος Πρέπει να τα αποφύγουμε αυτά βέβαια. Η δομή αποφασίζεται ανεξαρτήτως πριν από τις εκλογές και την δομή την καθορίζουμε μόνοι μας πριν τις εκλογές και πριν την παρουσίαση του περιεχομένου των χαρτοφυλακίων. Πάντα θα υπάρχει λοιπόν μια διαφορά μεταξύ των δύο αυτών. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να μην μακρηγόρησα και βαρεθήκατε για αυτό το εξαιρετικό έγγραφο. Ο Γιώργος Σέπλιν. Γιώργο! Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Εξαιρετική δουλειά και ο κύριος Πρέντα λίγο πολύ με κάλυψε, όχι όλα βέβαια, έχω κι εγώ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Και ήθελα να προσθέσω ότι νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, αλλάξαμε και την ημερομηνία των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πήγαν όλα νωρίτερα για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε μία νωρίτερη ημερομηνία. Δεν ξέρω αν η 1η Αυγούστου είναι η πλέον κατάλληλη, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει όπω ναι, καθυστέρησε, ναι. διότι και εγώ συμφωνώ ότι πιεστήκαμε πολύ από πλευρά χρόνου. Τώρα, για τι ακροάσει. Εγώ θεώρησα, και αυτό είπε και ο κύριο Πρέντα, ότι το να ακούσει έναν επίτροπο ε, τρεις ή και τέσσερις επιτροπές σε μια περίπτωση δεν είναι λογικό. Ούτως ή άλλως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει διαφάνεια, είναι να περάσουν οι επίτροποι από μια διαδικασία ε, ερωταποκρίσεων και να ε, δούμε τι γίνεται. Ε, και νομίζω ότι υπάρχει και το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος και δεν ξέρω αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα υπήρχε δυνατότητα επερωτήσεων. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, γιατί και πώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να ε, το συζητήσω πολύ το, το ζήτημα, αλλά τελικώ κάποιε από τι ακροάσει έγιναν ένα πολιτικό θέατρο. Κάνανε ερωτήσει, απαντούσαν οι επίτροποι και τέρμα. Και Ε, μείναμε ξεκρέμαστε λίγο, διότι κάποιοι από του επιτρόπους... Ε, έδωσαν τόσο τυποποιημένες απαντήσεις, τουλάχιστον σε αυτές που συμμετείχα εγώ, που πραγματικά ήταν ιδιαίτερα ενιαρή όλη η διαδικασία. Και δεν ε, θεωρώ ότι κάποιος τέθηκε υποδοκιμασία, τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, κυρίω όσον αφορά την παραβίαση από πλευρά τη διάσκεψη των Προέδρων ε, τη διαδικασία. Δεν ξέρω, είτε εσεί είτε ο κύριο Πρέντα ε, νομίζω ότι αν εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώ μιλάμε για το κράτο δικαίου, πρέπει τουλάχιστον να τηρούμε εμεί του κανόνε μα. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είναι δική σα μένει η έκθεση, αλλά εγώ πραγματικά θα ήμουν πιο αυστηρό, ε, στη διατύπωσή μου. Μπορεί να θέλετε να είστε πιο ήπιος, αλλά εγώ πραγματικά το έχω στην καρδιά μου το ζήτημα αυτό. Μετά, η παρατήρηση του κυρίου Πρέντα, πάλι, το διορθωτικό ζήτημα, όντως θα πρέπει να περιλαμβάνει και αυτή τη δυνατότητα ένας νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορεί πλήρως να αναδιαρθρώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό φυσικά θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη δική μας τη ζωή. Και αυτό συνέβη. Όταν το έθιξε αυτό στον κύριο Γιούγκερ, μου είπε είναι πρόβλημα του Κοινοβουλίου. Στην πραγματικότητα όμω δεν είναι πρόβλημα του Κοινοβουλίου, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τι ακροάσει μα μετά με ε, τον ίδιο βαθμό ε, ακρίβειας που θα θέλαμε. Και μια τελευταία παρατήρηση για τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι σε κάποιο σημείο η διαφάνεια γίνεται παραβίαση ε, ιδιωτικής ζωής και δεν ξέρω πού είναι η διαχωριστική γραμμή. Αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο προέκυψε το ζήτημα, κάποιος ο οποίος μεταβίβασε μετοχές σε μέλη τη οικογένεια του, αλλά σε ποιο σημείο γίνεται παρέμβαση των μελών τη οικογένεια, την προστασία των δικών του δεδομένων. Είναι δύσκολο το θέμα, υπάρχουν πολλέ πτυχέ. Νομίζω όμω ότι εγώ θα ήθελα να έχουμε λίγα περισσότερα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ η Mercedes Πρέσο. Ευχαριστώ. εγώ έχω μια παρατήρηση. Πρώτον, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, ε, e είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και μια ε, γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας και μετά να καθορίσουμε μετά από το κείμενο, ένα κείμενο συγκεκριμένο το οποίο θα κάνει κάποιες προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση και έχουμε τη δυνατότητα από εκεί και πέρα να τροποποιήσουμε και να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη πρόταση. Δεύτερον, και εγώ νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το χρόνο. Πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο τις διαδικασίες, γιατί η δική μας η Επιτροπή ιδίως πιέστηκε πάρα πολύ από την επιλογή της διάσκεψης των Προέδρων, διότι ε, περιορίστηκε πάρα πολύ η δυνατότητα συζήτησης με τον Τίμερμανς. Αλλά κυρίως θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο της διάσκεψης των Προέδρων και αυτό που επεσήμανε και ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ ε, όσον αφορά ερωτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να τίθεται στον κάθε επίτροπο, ακόμα και αν είναι ο αντιπρόεδρος αυτός, αλλά μπορούν να τίθεται μόνο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια άτυπη, ανεπίσημη ε, ακρόαση, διότι είναι σαφές, διότι δεν ε, περνάει από ακρόαση ο πρόεδρος επισήμως, αλλά είναι μια ε, ανεπίσημη ακρόαση στην οποία διευκρινίζει κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να διευκρινίσει ο κάθε επίτροπος, διότι πραγματικά τη νιώσαμε αυτή την ανάγκη με αυτή τη νέα διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου οι αρμοδιότητες είναι λίγο πιο ρευστές και φυσικά υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο συντονισμού από πλευράς Προέδρου ακριβώς λόγω αυτού. Θεωρώ ότι μια πρώτη πρόταση είναι αυτή της αξιολόγησης, θα πρέπει να το επεξεργαστούμε, αλλά όντως ε, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τις αξιολογήσεις. Αν γίνουν κατά τρόπον ώστε να μην φτάνει κάποιος αμέσως σε ψηφοφορία, αλλά αν υπάρχει κάποια στάδια στο ενδιάμεσο θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, Θεωρώ ότι όντως πρέπει να επισημοποιήσουμε σε γνωμοδότηση τουλάχιστον την πρόταση ε, για δύο τουλάχιστον υποψηφίου. Θα δούμε στη συνέχεια αν θα είναι δύο ή τρει, ώστε να υπάρχει και ίση εκπροσώπηση φύλων, χωρί να υποχρεώνονται οι χώρε οι οποίε έρχονται τελευταίε να διορίσουν γυναίκε, γιατί αλλιώ ε, δεν βγαίνουν τα νούμερα και δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε, γιατί δεν είναι και δίκαιο αυτό. Αν και ε, αφού καθυστέρησαν, κάπου πρέπει να λάβουν και τι ευθύνε του. Αλλά δεν είναι πολύ δίκιο, αλλά και επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ ε, κυβερνήσει συνασπισμού πλέον, το να διορίσει κάποιο τρεις ε, υποψηφίου, θα επέτρεπε και στον ε, πρόεδρο να έχει καλύτερη εκπροσώπηση και βάσει κυβερνήσεων των χωρών και βάσει Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει σημασία λοιπόν και για ισορροπία λογοφύλων αλλά και ισορροπία λόγω πολιτικών δυνάμεων. Δεν θα επισέλθω τώρα στην ουσία κάποιων άλλων σημείων. Θα το κάνουμε αν υπάρξει δυνατότητα για γνωμοδότηση. Νομίζω ότι θα το θέσει η πρόεδρος στην ημερήσια διάταξη και να αποφασίσουμε ή θα μπει στον κανονισμό στην ομάδα εργασίας αυτή ή θα υπάρξει μια ad hoc γνωμοδότηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμη μια ad hoc γνωμοδότηση διότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ε, είναι αυτούσιο. Επομένως, αν ε, αυτούσιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλύτερη συζήτηση με όλο το Κοινοβούλιο και με τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ρίτσαρτ, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και μας έδωσε τη δυνατότητα και να συζητήσουμε το ζήτημα και τροφή για σκέψη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να, παρουσια... να υπενθυμίσω εδώ πέρα την απόφαση των μη εγγεγραμμένων μελών για την διαδικασία αυτή. Αντιλαμβάνομαι πως οπωσδήποτε θέλετε να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών που είναι ενταγμένοι σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα και αυτών που δεν είναι και αντιλαμβάνομαι πως η διαδικασία λήψη αποφάσεων όσον αφορά τους ε, επιτρόπους δεν θα κριθεί από τα μη ενταγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ουδέτερο και έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να σχηματίσει μία άποψη και να μην περιοριστούμε σε, στους βουλευτές μόνο ε, που είναι μέλη ε, μια συμβουλευτική ομάδα ή μια επιτροπή. Θα πρέπει να γίνεται ο συντονισμό τουλάχιστον με του ε, συντονιστέ για να έχουμε και εμεί την δυνατότητα να μιλήσουμε, να εκφραστούμε σε σχέση με του επιτρόπου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Durand. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω πολύ αλλά δεν ήθελα να ξεχάσουμε ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον κύριο Κόρμπετ για όλη του τη δουλειά. Η έκθεσή του είναι σαφέστατη και προσπαθεί να ταυτίσει όντως αληθινά θέματα λέγοντας ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες. Και εγώ είμαι καινούριο βουλευτής και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι και έγγραφα γιατί έτσι προχωράμε. Είναι θέμα αρχής βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Δεύτερον, εμένα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα των φύλων αλλά και της πολιτικής εξισορρόπησης. Πρέπει να σεβόμαστε την πολιτική εξισορρόπηση, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί αν κάποιος είναι άντρας ή γυναίκα να βλαφθεί, να ζημιωθεί αυτή η πολιτική εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση των φίλων γίνεται σε πολλά κοινοβούλια και μπορεί να επιτρέψει, ούτως ή άλλως είμαστε υποχρεωμένοι, να καταλήξουμε στην ισότητα. Αυτό θέλουμε όλοι. Βέβαια δεν είναι προβλήματα όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε, αλλά υπάρχει θεωρία, υπάρχει και πρακτική. Εμείς τις ε, αυτές διαπιστώσαμε ότι υπάρχει θέμα ισορροπίας που μειώνει τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου να συζητήσει πραγματικά για τις ικανότητες ορισμένων επιτρόπων. Εγώ είδα κρόάσεις κυρίως του κυρίου Μοσκοβισή μετά του κυρίου Κανιέτε ότι ήταν ένα παιχνίδι της εξουσίας και είναι πολύ δύσκολο για έναν κοινοβουλευτικό που θέλει να είναι αντικειμενικός και να δει αν ο Α ή ο Β επίτροπος είναι ο ικανότερος, είναι πολύ δύσκολο να βλέπει να καταστρέφεται η ισορροπία από τις συμφωνίες μεταξύ ομάδων. Υπάρχει εδώ ένα θέμα, το οποίο ίσως να μην έχω απάντηση, αλλά το Κοινοβούλιο δεν ωφελείται νομίζω από τέτοιου είδους συμφωνίες διαδρομιστικές και ούτε οι πολίτες τα εκτιμούν όλα αυτά ιδιαίτερως. Και τώρα κάτι άλλο για τις διαμάχες μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων και τα, τις δηλώσεις συμφερόντων. Αυτό είναι υποχρεωτικό, αλλά το νομικό πρόβλημα που τίθεται είναι ότι εξετάζουμε μόνο τα άμεσα συμφέροντα ενώ για τις δικαιοδοσίες τους για το χαρτοφυλάκιο αυτά τα εξετάζει μόνο η Κομισιόν. Υπάρχει εδώ λοιπόν μία διαφορά. Ή δεν θα μιλήσουμε καθόλου για τα οικογενειακά συμφέροντα ή θα το λέμε συνέχεια, αλλά όχι αυτή την ανισορροπία μεταξύ της δήλωσης που εξετάζει το Κοινοβούλιο και της δήλωσης που εξετάζει η Κομισιόν. Είναι θέμα ισότητας και αυτό. Και τέλος, ξέχασα τι ήθελα να πω τελευταίος, δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Ευχαριστώ ο κύριος Χαστάλδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κόρμπετ για τη δουλειά του. Η έκθεσή του είναι πολύ σαφής και εξονυχιστική. Συμφωνώ με τον κύριο Ντουράν ότι ίσως δεν είναι καλή ιδέα να γίνονται πάντοτε αυτά τα παιχνιδάκια ισορρόπησης, εξισορρόπησης μεταξύ των πολιτικών ομάδων γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί κανέναν, είναι μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων ομάδων. Και ελπίζω στο εξή να γίνει εξαίρεση και όχι κανόνας. Γιατί αλλιώς θα σήμαινε ότι δεν κάνουμε αντικειμενική ανάλυση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Απλώς παίζουμε ρόλους και κάτι που με ενόχλησε ιδιαίτερα κατά τις ακροάσεις αυτές ήταν η ακρόαση του κυρίου Τίμερμανς όπου εφαρμόστηκε τελείως εξαιρετική διαδικασία σε σύγκριση με τον αλλονόν. και θα ήθελα να συνεργαστούμε ώστε να συμφωνήσουμε για αυτά τα θέματα να είναι επαναλαμβάνω εξαίρεση και όχι κανόνα αυτά τα παιχνίδια όλοι οι επίτροποι και οι αντιπρόεδροι της Επιτροπής και οι πρώτοι αντιπρόεδροι και όλοι όλοι μου φαίνεται ότι είναι σωστό να ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και ιδίως στις διεθνείς σχέσεις η ύπαρξη των κλάστερ φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει για θέματα πολιτικών εξωτερικών σχέσεων και εμπορικών ακόμη σχέσεων. Όχι Παναγία Και ελπίζω ότι η διαδικασία δεν θα, ξανά, δεν θα επαναληφθεί ξαν, ποτέ ξανά. Δεν θα επαναληφθεί. Σας ευχαριστώ. Ρίτσαρτ, δυόμιση λεπτά Σύντομα. Ναι. Σύντομα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο και σε γενικέ γραμμές νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο βαθμό συνένεση για διάφορα θέματα. Βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα των ερωτήσεων και του είδους των ερωτήσεων Ε, κάποια ομάδα, δεν ξέρω η μέλος, διαφώνησε από αυτού είπα σαφέστατα για τις επερωτήσεις ότι ήταν κατά των κανόνων αυτό, επομένως θα πρέπει να αποφασίσουμε ή θα αλλάξουμε τους κανόνες ή θα τους πούμε μην το ξανακάνετε. Δεν ξανακάνετε. Για τη διάσκεψη των Προέδρων βέβαια μέχρι τότε θα έχουμε καινούργια, οπότε θα δούμε. Για τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, ναι, όντω είναι λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ διαφάνειας και ε, παραβίασης προσωπικής ζωής Πάντα έτσι γίνεται με αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Ντουράν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Να δούμε τη διαφορά που ήδη υπάρχει. Ναι, θα το σκεφτώ για τον κύριο Χάνεμανς. Εγώ δεν μπορώ να πω συλλογικά τι άποψη έχουν οι συνάδελφοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Ντουρόμ, σας ευχαριστώ πολύ. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Ένα μόνο. Για αυτά τα παιχνίδια των πολιτικών ομάδων που κρατούν ομήρους ο ένας τον άλλον, ε, εδώ είναι πολιτικό κοινοβούλιο. Σαφώς και οι πολιτικές αξιολογήσεις μπορεί να επηρεάσουν την κρίση κάποιων. Αν πραγματικά όμω οι πολιτικέ ομάδε ήταν αυστηρά και έλεγαν ότι θα υποστηρίξουμε μόνο του δικού μα, δεν θα είχε περάσει ούτε ένα επίτροπο. Σε γενικέ γραμμέ οι ομάδε ήταν διατεθειμένε να δεχτούν ο ένα τι υποψηφίου των άλλων. Αλλά υπάρχει και μια δικλίδα ασφαλεία εδώ για να ξεφορτωθούμε έναν Επίτροπε που το κάναμε και τώρα και την προηγούμενη φορά και λοιπά. Ε, δεν έχει νομική βάση, αυτό είναι πολιτικό. Τα καταφέρνουμε μόνο όταν υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση και ε, η κυριαρχία απόψε ότι δεν ήταν καλός ο επίτροπος. Αν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, δηλαδή κάθε φορά λέμε ότι να αλλάξει αυτόν και εκείνον και τον άλλο και αλλάζουμε τη μισή επιτροπή, νομίζω ότι ε, ουσιαστικά δεν θα, μπορούμε, θα παραλύσουν τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία λοιπόν και η ισορροπία ακριβώς είναι αυτό το πάρε δώσε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ναι, έχουν την τάση οι ε, ομάδες να επιτίθενται το ένα στον επίτροπο του άλλου, αλλά όχι ε, επιθετικά, γιατί αλλιώς ε, δεν ε, θα λειτουργούσαν τα πράγματα. Θα το ξαναδούμε. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση. Το ξέρετε κυρία Πρόεδρε ότι θα πάω και στην ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών για να ακούσω και τις δικές τους απόψεις από τους διαφόρους Προέδρους που προείδρευσαν στις ακροάσεις. Ο Φραν Τίμερμανς μου υποσχέθηκε τουλάχιστον ανεπίσημα ότι θα μου εξηγήσει και την άποψη των Επιτρόπων πώς το είδαν αυτοί το ζήτημα. Ε, και έχουμε λοιπόν και κάποιες άλλες πληροφορίες από αυτούς και φυσικά δεν υπάρχει λόγος βέβαια να διαβιαστούμε, αλλά εν ευθέτω χρόνο θα μπορούσαμε κάλλιστα αυτό να το κάνουμε ένα σχέδιο έκθεσης ε, υπομορφή ψηφίσματος ενδεχομένως για το Κοινοβούλιο το οποίο σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να ζητήσει και αλλαγή του κανονισμού και σε κάποια άλλη παράγραφο μπορεί να λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το ΤΑΔΕ με την Επιτροπή ή με το Συμβούλιο και σε μια άλλη παράγραφο να λέει ότι καταλήγουμε στο ΤΑΔΕ συμπέρασμα για το Κοινοβούλιο για την επόμενη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι επόμενε ακροάσει. Ανάλογα με τη μορφή των συμπερασμάτων, κάποια από αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω και να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία, όπω για παράδειγμα η γενικότερη αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων, ε, που ελπίζω να επιφολήθηκαν και από τη συζήτηση για τις ακροάσεις, ε, για τις δικές τους εργασίες. Η ΑΦΚΟ ζήτησε μία μελέτη για να εξετάσει λίγο καλύτερα τη διαδικασία των ε, ε, ευρωπαϊκών κομμάτων ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ έχουμε μια μελέτη από του εμπειρογνώμονε που είναι εδώ μαζί μα, ο καθηγητή Λουτσιάνο Μπάτζε από το Πανεπιστήμιο τη Πίζα, επίση και ο καθηγητή Εουτζένιο Πιτσιμέντη και από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο τον δόκτωρα Ερίκο Καλώση και τον κύριο Γκαγκάτεκ από το Κέντρο για την Ευρώπη του Πανεπιστήμιου της Βαρσοβίας. Εσείς θα διοργανώσετε ποιος θα μιλήσει πότε. Έχετε το ε, λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσίαση αυτή λέγεται πολιτικά κόμματα και ιδρύματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο προκλήσεις και ευκαιρίες. Δύο από τους συντάκτες είναι εδώ. Ο Εντουάρτε Περσίνελη και ο Λορέντζο Τσίκη. Λοιπόν, πώς έχει η παρουσίαση. Μία εισαγωγή και τρία μέρη. Η θέση πολιτικής και η συνοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομάδων μετά την Ευρωκρίση, η ρύθμιση και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη αυτή βασίζεται, είναι συνέχεια βασικά μιας προηγούμενης μελέτης για το πώς να δημιουργηθεί ένα υπερεθνικό σύστημα κομμάτων που επίσης μας είχε αναθέσει η ΑΦΚΟ το 2010 από το Παρατηρητήριο Πολιτικών Κομμάτων όπου έγινε και αυτή η μελέτη. Η αρχική μελέτη έβλεπε τα πολιτικά κόμματα και το δόγμα του στο πλαίσιο μιας σύγκλησης εντός των πολιτικών ομάδων του ΕΛΚ. Η συνοχή λοιπόν όσον αφορά τις ε, ψηφοφορίες και η σύγκληση εντός αυτών των ομάδων και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα πολιτικά κόμματα για να επιλέξουν υποψηφίους ε, για τις ευρωεκλογές. Το άλλο ήταν πώς θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός ε, ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικών κομμάτων που ήταν η ουσία της μελέτης εκείνης και τέλος προτάσεις για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού συστήματος και των συστημάτων χρηματοδότησης των κομμάτων. Η μελέτη έτυχε θερμής υποδοχής ε, στον πανεπιστημιακό χώρο, έγιναν πολλές παραπομπές σε αυτήν, οπότε ευχαριστούμε την Επιτροπή σας, αλλά προφανώς ε, έτυχε θερμής υποδοχής και εδώ μέσα, καθώς μας ζήτησαν ε, συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες διαφορές με την τωρινή μελέτη, γιατί η τωρινή δεν περιλαμβάνει δύο πτυχές που είχαμε καλύψει το 2010. πρώτη αφορά τις διαδικασίες επιλογής ε, υποψηφίων ευρωβουλευτών. Και αυτό, αντιλαμβανόμαστε, είναι αντικείμενο μιας άλλης μελέτης που επίσης ζήτησε η ΑΦΚΟ. Η άλλη πτυχή που δεν καλύψαμε είναι ο εκλογικός νόμος. Α, μάλιστα, ναι. Με συγχωρείτε. Ξέχασα να πατήσω το κουμπάκι. Ε, το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Το συζήτησαν δηλαδή άλλοι εμπειρογνώμονες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα τα θίξουμε αυτά τα θέματα. Θα το κάνουμε στις ε, συστάσεις μας. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα ουσίας ε, θέσεις ε, και συνοχή των ε, πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την Ευρωκρίση. Εμείς αναλύουμε εδώ πέρα τις θέσεις και το επίπεδο συνοχής στις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του να εστιάζουμε στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσεις ε, στις πιθανές διαφορές εντός των ομάδων αυτών. Τι εννοούμε δηλαδή. Υπήρχε η ανησυχία πως θα, θα επηρεαστεί η εσωτερική σύνοχη των α, κοινοβουλευτικών ομάδων. Και μια απόκληση μεταξύ των αδελφών κομμάτων και έτσι ότι θα έχουμε μια νέα εδαφική Δευκό διαχωρισμό μεταξύ ευρωβουλευτών από τα βόρεια και τα νότια κράτη-μέλη. Όπως είπα, ήταν σοβαρή αυτή η ανησυχία και θεωρούσαμε πως έπρεπε να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Χρησιμοποίησαμε τρεις διαφορετικές πηγές δεδομένων. Το ευρωβαρόμετρο, τις ε, έρευνες ε, σε βουλευτές που έκαναν εδώ και χρόνια διάφοροι πανεπιστημιακοί και μετά βεβαίω τα δεδομένα από τις ονομαστικές ψηφοφορίες. Ποια είναι τα ευρήματα. Τα ευρήματα είναι θετικά Όπως μας δείχνει το ευρωβαρόμετρο, οι διαφορές μεταξύ βορείων και νοτίων κρατών μελών παραμένουν μικρές και δεν έχουν αυξηθεί μετά την κρίση. Μισή έκπληξη, αλλά αυτό λένε τα δεδομένα. Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκε κάποια κάποιος εδαφικός διαχωρισμός και ιδιαίτερα σημαντικό ήταν αυτό σε σχέση με τις ε, ονομαστικές ε, ψηφοφορίες. Αλλά επίσης αυτό φάνηκε και από τη στάση των βουλευτών με βάση τις συνεντεύξεις τους, κάτι το οποίο βεβαίως δεν θα φαινόταν στην ψηφοφορία λόγω της κομματικής πειθαρχίας. Άρα τα συμπεράσματα είναι αισιόδοξα για το ευρωπαϊκό σύστημα κομμάτων και δεν θεωρούμε ότι έχει επηρεαστεί από την κρίση. Το τονίζουμε αυτό γιατί η συνοχή και η σύγκληση εντός των ομάδων ιστορικά είναι ε, ένα ισχυρό σημείο του ευρωπαϊκού κομματικού συστήματος. Οπότε το ότι δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί, ε, προφανώς οι ευρωεκλογέ του 2014 είχαν κάποια αποτελέσματα, αλλά όχι ε, εντός των ομάδων. Και περνάμε στο επόμενο τμήμα και σβήνει το μικρόφωνο. Θα σας το παρουσιάσει ο Εουτζένιο. Θα παρουσιάσω σύντομα τις ε, βασικές θεωρητικές υποθέσεις της μελέτης μας για τον αντίκτυπο της ρύθμισης και χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως ένα καθεστώς ρύθμισης και χρηματοδότησης βοηθούν στην θεσμοποίηση των κομμάτων και των κομματικών συστημάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μη σταθεροποιημένα πολιτικά συστήματα όπου το κράτος ευνοεί τα πολιτικά κόμματα για να αυξηθεί η ποιότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αλλά η διαδικασία αυτή κρατικοποίησης ας πούμε αποκαλύπτει και μια αλλαγή στην φύση τους από ιδιωτικές ενώσεις που δημιουργήθηκαν για να εκφράσουν συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνίας, τα κόμματα έγιναν ένα περίεργο είδος δέκο με κύριο στόχο να συνεισφέρουν στην παραγωγή συλλογικών αγαθών μέσω του ρόλου τους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. δηλαδή λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και άρα και το κράτος έχει δικαίωμα να ρυθμίσει τις δραστηριότητες τους. Βλέπουμε εδώ πέρα τι συνέβη 10 χρόνια μετά την ε, εισαγωγή του συστήματος αυτού το 2003-2004 και μετά την υιοθέτηση του νέου κανονισμού. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση συγκρίνουμε την χρηματοδότηση σε κράτη-μέλη και μετά το εφαρμόζουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε δύο διαστάσεις και τέσσερις υποδιαστάσεις για την κάθε μία. Θα τα πούμε μετά. Οπότε οι βασικές ελλείψεις του κανονισμού 2004-2003 ήταν τουλάχιστον τρεις. Πρώτα απ' όλα ήταν μια σειρά κανόνων που όριζαν τη χρηματοδότηση αλλά δεν αναφέρθηκε σε βάθος στο ζήτημα της ε, οργανωτικής εδραίωσης των κομμάτων. Κατόπιν ήταν υπέρ της υπαγωγής των ευρωπαϊκών κομμάτων στα εθνικά και ειδικά στην ε, φάση αυτή την θεσμική καθώς τα κονδύλια τα διαχειριζόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τρίτο και σημαντικότερο δεν άνοιγε το βασικό ζήτημα. Πώς θα συνδεθούν τα ευρωκόμματα με τους Ευρωπαίους πολίτες. Μετά από 9 χρόνια η έκθεση Γιαννάκου και η σχετική ε, πρόταση της Κομισιόν είχαν στόχο να ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ ευρωκομμάτων και Ευρωπαίων πολιτών. Αφενός, προωθώντας τη διαδικασία μιας οργανωτικής σύγκλησης ε, μέσω ε, κάποιων αυστηρότερων προϋποθέσεων για πρόσβαση σε δημοσία κονδύλια. Από την άλλη, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές όπως αυτές που αφορούσαν ε, το πώς γίνεται κανείς μέλος του κόμματος και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Όμως το σχέδιο κανονισμού που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Τα ευρωπαϊκά κόμματα συνεχίζουν να ε, αντλούν κυρίως δημόσια κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν χαλαρώσει τα όρια για την ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά είναι υψηλότερα από αυτά που πρότεινε η έκθεση Γιαννάκου. Η απαγόρευση για χρηματοδότηση των εθνικών κομμάτων δεν βοηθάνε στο να μάθει ακόμα και την ύπαρξη των ευρωκομμάτων ο Ευρωπαίος πολίτης. Οπότε είναι κατά την άποψή μας πρόωρο να μιλήσουμε για ένα σύστημα ε, ευρωπαϊκών κομμάτων ή ευρωπαϊκή αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Καθώς ε, αυτό δεν θα γίνει μέχρι να ενισχυθεί ο ρόλος του σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα ή μια ευρωπαϊκή πόλη. Okay, thank you very much. And we would like now to... Θα θέλαμε τώρα να περάσουμε στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης μας, το ρόλο των πολιτικών ιδρυμάτων. Η έκθεση του 10 που ανέφεραν μερικοί δεν εξέτασε το ρόλο των πολιτικών ιδρυμάτων διότι η αναπτύξη τους τότε ήταν ακόμη εμβριακή. Αλλά τα επόμενα χρόνια συνέχισαν τις δραστηριότητες τους, αυξήθηκαν αυτές και γι' αυτό αποφασίσαμε να τα συμπεριλάβουμε. Θα μπορούσε κανείς να αναμένει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναλύσει κανείς τη δραστηριότητά τους, αλλά εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον δικό μας, τη σύνδεση δηλαδή των ευρωιδρυμάτων με τα ευρωπαϊκά παλιτικά κόμματα. Θα ήθελα καταρχήν να σας εξηγήσω γιατί είναι έτσι η φύση αυτής της σύνδεσης ευρωκομμάτων και ευρωιδρυμάτων που θα μπορούσε να είναι σημαντικός παράγον για την αναπτύξη ε, διακομματικών ψυχοδελτίων. Ένα λειτουργικό κομματικό σύστημα απαιτεί ορισμένες δομημένες σχέσεις μεταξύ κομμάτων που να βασίζεται σε πολιτικό ανταγωνισμό για την βέβαια. Πέρα από τις εκλογές και τον ανταγωνισμό αυτό τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να βασίζονται σε μια προγραμματική βάση. Και σε αντίθεση με τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ευρωκόμματα δεν έχουν αρκετούς υλικούς πόρους και προσωπικό για να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους και γι' αυτόν τον λόγο η ίδρυση ευρωιδρυμάτων τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες ιδέες, να γίνουν πιο λειτουργικά. Παρ' όλα αυτά, και θα ήθελα αυτό να το τονίσω ιδιαίτερα, αυτή η σύνδεση με την εμφάνιση των ευρωιδρυμάτων και την αναπτύξη ε, διενοσιακών ε, κομμάτων δείχνει ότι δείχνει ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός τους ρόλος. Αυτό είναι και το ερώτημα που θέτουμε και που βλέπετε εδώ στην διαφάνειά μας. Σε αυτό το τμήμα της έκθεσης χρησιμοποίησαμε τρεις πηγές δεδομένων. Την ακαδημαϊκή φιλολογία και τα αποτελέσματα μίας διάσκεψης που συνδιοργανώσαμε με την ΑΦΚΟ το 2013 και όπου ήρθαν εκπρόσωποι πολλών ευρωιδρυμάτων καθώς και τη μελέτη του Ιανουαρίου 2014. Και παρά την συσσόρευση αυτή εμπειρικών στοιχείων θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ακόμα είμαστε στη φάση της διαπίστωσης. Χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση για να δούμε τα πράγματα σφαιρικότερα για το ρόλο των Ιδρυμάτων. Και στην παρουσίασή μας θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Επειδή δεν υπάρχει πολύς χρόνος θα ήθελα εδώ να περιοριστώ σε στοιχειώδη στη, ε, δεδομένα. Όπως ποιος ελέγχει τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των ευρωιδρυμάτων. Πρώτον με τη χρηματοδότηση. Λόγω της πολιτικής οργάνωσης του Κοινοβουλίου, οι μεγαλύτερα δύο ευρωιδρύματα είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, που τώρα λέγεται Wilfried Mertens, που σχετίζεται με το ΕΛΚ, και το Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Προόδο των σοσιαλιστών. Αυτά είναι τα κύρια και τα, αυτά που αφοροφούν τα περισσότερα χρήματα. Με βάση τις πόρους τους του 2014, το κέντρο Wilfried Mertens έλαβε 4,2 δισεκατομμύρια, 34% δηλαδή του συνολικού, του, του συνολικού προπολογισμού των ευρωιδρυμάτων και το άλλο των σοσιαλιστών 2,8 δισεκατομμύρια, 24% τα μικρότερα ιδρύματα όπως η οργάνωση για την διακρατική συνεργασία στην Ευρώπη 107.000 περίπου ευρώ δηλαδή 1,4% του συνολικού προϋπολογισμού για τα Ιδρύματα. Θέλουμε να τονίσουμε λοιπόν ότι αυτό το μεγάλο χάσμα μεταξύ των πόρων που χορηγούνται εξηγεί πολλές από τις διαφορές των Ιδρυμάτων που θα σας δείξουμε σε λίγο. Ακόμη και αν όμως η αριθμοί αυτή είναι χαμηλή, πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πραγματικά τους πλαίσια. Λόγω της μικρότερης χρηματοδότησης που δίνεται στα μικρά ιδρύματα, παρά μάλλον το μικρό αυτό ύψος, μπορούν να συμπληρώσουν χρήσιμα τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων στην Ένωση και τα μεγάλα ιδρύματα δεν έχουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι προϋπολογισμοί δηλαδή των ιδρυμάτων είναι μεταξύ 64 και 70% του συνολικού προϋπολογισμού των πολιτικών κομμάτων στα, με τα οποία συνδέονται τα ευρωιδρύματα. Οι αριθμοί λοιπόν αυτή και το χάσμα δεν προδικάζει τη χρησιμότητα των ιδρυμάτων για τα πολιτικά τους κόμματα αν και επηρεάζεται βέβαια η χρηματοδότηση από τον αριθμό δραστηριοτήτων που μπορούν να αναλάβουν. Ανακαλύψαμε μεγάλες διαφορές μεταξύ μεγάλων και μικρών ιδρυμάτων και αυτό δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τον αριθμό των δημοσιεύσεων ή δραστηριοτήτων αλλά επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και στη φύση των σχέσεων που έχουν με τα αντίστοιχα τους κόμματα. Τα δύο μεγαλύτερα ευρωιδρύματα, ο Wilfrid Μέρτενς δηλαδή και το Ίδρυμα για το Ευρωπαϊκή Πρόοδο του ΕΛΚ και του Σοσιαστών, όπως είπα και προηγουμένως έχουν ισχυρότερους δεσμούς με τα ανάλογα κόμματά τους από ότι τα άλλα ιδρύματα με τα άλλα κόμματά τους. Και αυτές οι στερινότεροι δεσμοί φαίνονται και δυναμικά, στατικά και δυναμικά. Στατικά αυτό φαίνεται από την ανάλυση της σύνθεσης και των δικαιωμάτων ψήφου. Δηλαδή, στο Προεδρείο του ΦΕΠΣ, που αποτελείται από 20 μέλη, 6 από αντιπροσωπεύουν εθνικά think tank, ενώ άλλα 6 μέλη του κόμματος. Πολλές φορές τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιδρυμάτων είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου των Κομμάτων μέλη. Από δυναμικής απόψεως όμως, και μιλάω για το κέντρο Βιλπριμέρτεν και το κέντρο για το Ευρωπαϊκή Πρόοδο, οργανώνουν και δραστηριότητες μαζί με τα πολιτικά των κόμματα. Ιδιαίτερα τη συγγραφή του, μανιφέστου, του προεκλογικού μανιφέστου Υπάρχει όμως και άλλο πρότυπο ιδρύματος που δεν λειτουργεί έτσι. Τα μικρότερα ιδρύματα έχουν χαλαρότερους δεσμούς με τα κόμματά τους ως προς την κοινή σύνθεση των διοικητικών του συμβουλίων. Έχουν όμως και κοινέ δραστηριότητες. Ναι, ευχαριστώ Βόιτσεκ. Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο ήδη ανέφερε ο Βόιτσεκ τη δραστηριότητα των πολιτικών ειδημάτων, αλλά θα ήθελα να σας πω και λίγο καλύτερα τι θα έπρεπε να κάνουν βάσει της μελέτης. Βάσει της πλήρους εκδοχής του κανονισμού του 2004-2003, τα πολιτικά ιδρύματα, όπως βλέπετε και εδώ στη μελέτη μας, θα πρέπει να παρακολουθούν, να αναλύουν και να συνεισφέρουν στη συζήτηση για ευρωπαϊκά ε, θέματα δημόσιας πολιτικής και να, ε, τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, να αναπτύξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα ευρωπαϊκής ε, δημόσιας πολιτικής, όπως διοργάνωση ε, σεμιναρίων, επιμόρφωσης, διασκέψεων και μελετών και θέματα σχετικά, ε, σχέσεις μεταξύ ε, ε, ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και οργανώσει της νεολαίας και εκπροσώπους τη κοινωνίας των πολιτών. Επίση, θα πρέπει να αξιολογούν ε, την ανάπτυξη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς προκειμένου να προωθήσουν τη δημοκρατία και τέλος η σχέση μεταξύ τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και τα εθνικά πολιτικά ιδρύματα. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποτελούν το πλαίσιο για τα εθνικά πολιτικά ιδρύματα, για τον ακαδημαϊκό κλάδο και άλλους ε, σχετικούς φορείς σε συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι στη μελέτη. Αυτά τα έχουμε στο χαρτί. Τι έγινε στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε το πραγματικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας των ε, Ιδρυμάτων. Έχουμε χωρίσει τις δραστηριότητες ανά έτος. Θεωρούμε ότι είναι οι συνήθεις δραστηριότητες αυτές που γίνονται στη διάρκεια του μια συνήθους χρονιάς και από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε και σε ειδικέ χρονιές, για παράδειγμα ε, τη χρονιά των ευρωεκλογών. Αυτή είναι η ειδική χρονιά. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν στις συνήθεις δραστηριότητες τους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διοργανώνουν εκδηλώσεις, και αν θέλετε να το διαβάσετε στο έγγραφό μας θα δείτε ότι υπάρχει και βαθμολόγηση των διαφόρων πολιτικών ιδρυμάτων ανάλογα ε, με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν και θα δείτε ότι το 2013 κάποιες οργανώσεις δεν οργάνωσαν τίποτα, κάποια ιδρύματα συγγνώμη δεν οργάνωσαν τίποτα, ενώ κάποια άλλα ιδρύματα διοργάνωσαν 54 εκδηλώσει. Από το 0 έως το 54 έχουμε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα τα οποία κυμαίνονται εδώ μέσα. Το άλλο σημαντικό αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων είναι οι δημοσιεύσει του. Και υπάρχουν διάφορε μορφέ δημοσιεύσεων. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα. Αυτό είναι μια μορφή ε, δημοσιοποίηση στοιχείων. Ε, ένα περιοδικό ή αρκετά περιοδικά, βιβλία, ερευνητικές μελέτες, ή, ε, μελέτες πολιτικής ή διάφορες άλλες δημοσιεύσεις και υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται τώρα στη διάρκεια των εξαιρετικών ετών. Ε, ζητήσαμε τους υπαλλήλους του Euro των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, τι σκοπεύουν να κάνουν εν ώψη των ευρωεκλογών. Κάποια πολιτικά ιδρύματα διοργάνωσαν κάποιες ειδικέ εκδηλώσεις για να ε, εκπαιδεύσουν εθελοντές για τις προεκλογικές εκστρατείες ή και πιθανούς υποψηφίους. Κάτι ακόμα που σημαίνει ότι δεν διοργάνωσαν όλα τα ε, πολιτικά ιδρύματα ειδικέ εκδηλώσεις για κατάρτιση υποψηφίων, τι έγινε ε, ε, με το μανιφέστο των πολιτικών κομμάτων. Κάποια πολιτικά ιδρύματα δηλώνουν ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ε, κατάρτιση του εκλογικού μανιφέστο της, του αντίστοιχου πολιτικού τους κόμματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να πω και δύο λόγια παραπάνω για δύο πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν και σήμερα το πρωί κυρίως ε, η πρωτοβουλία των πολιτών και η πρόταση για ε, ένα πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Εδώ θα κλείσω τις διαφάνειες. Όπως είπε και ο καθηγητής ε, Μπάρντι, η μελέτη μας είναι συνέχεια της προηγούμενης μελέτης του 2010 που είχε τίτλο «Πώς να δημιουργήσουμε ένα πολυεθνικό σύστημα κομμάτων» είναι σημαντικό αυτό, αλλά είναι σημαντικό να ε, επανέλθουμε και στην αρχική μας έκθεση του 2010. Να σας πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Το 2010 εμείς στην έκθεσή μας ε, προτείναμε σαφέστατα ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ε, διαδικασίες των πολιτών και μέχρι τώρα τα πολιτικά κόμματα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο ε, ή είναι μηδαμινός ο ρόλος τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ειναι μηταμινός ο ρολος Συνταγματικών Υποθέσεων θα μπορούσε να υπενθυμίσει ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να διαδραματίζουν αυτό το ρόλο στην πρωτοβουλία των πολιτών. Και δύο λόγια για τον... Ε, αυτή τη, το ψηφοδέλτιο το πανευρωπαϊκό, το ψηφοδέλτιο επικρατείας αν θέλετε. Σήμερα ακούστηκε ότι ίσως δεν θα γνωρίζουμε αυτούς τους 25 υποψηφίους που θα είχαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και σε εθνικό επίπεδο. Οι ψηφοφόροι συνήθως δεν γνωρίζουν τους υποψηφίους των, των κομμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι οι επικεφαλής, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, οι επικεφαλής της λίστας. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την πανευρωπαϊκή λίστα, τουλάχιστον οι ψηφοφόροι θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουν ε, ε, τα ονόματα ή την ε, σταδιοδρομία των υποψηφίων, θα ξέρουν ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα. Και αυτό είναι καλό, θεωρούμε. Uh, Μία σύσταση τώρα, η οποία σχετίζεται και με την πρωινή συζήτηση. Ένας συνάδελφος Αναφέρθηκε ήδη στην ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα δεν μπορούν στις μέρες μας να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διάρκεια των εθνικών ε, εκλογικών προεκλογικών εξερατών. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πιο χαλαρά ε, όρια για τα ευρωπαϊκά κόμματα, διότι εμείς θεωρούμε ότι η πολιτικοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου θα μπορούσε να περνάει και από τον εξευρωπαϊσμό των εθνικών προεκλογικών εξερατιών. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις για τις επιστημονικές συστάσεις για περαιτέρω έρευνα. One is about foundation. Ένα πράγμα για τα πολιτικά ιδράματα. Ε, ο Βόιτσεκ έκανε μια πολύ καλή ανάλυση και έκανε ένα συσχετισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Λόγω έλλειψη χρόνου και χώρου στην έκθεση δεν εξετάσαμε τι σχέσει μεταξύ εθνικών πολιτικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η στάση, ο προσανατολισμό και οι προσδοκίε των μελών των εθνικών πολιτικών ιδρυμάτων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Αυτό είναι ένα περαιτέρω σημείο περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης. Και δεύτερον, ε, εκλογική νόμη. Σήμερα αναφέρθηκε η σημασία της διαφοράς ε, ε συστήματος ανοιχτού ψηφοδελτίου και λίστας. Και το σκεπτικό ήταν ότι το να υπάρχει ένα ανοιχτό ψηφοδέλτιο θα μπορούσε ίσως να είναι σημαντικό προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις, στις εκλογές. Στο παρελθόν, οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν υπάρχει ένα ανοιχτό ψηφοδέλτιο, αντί να αυξάνεται η συμμετοχή, επηρεάζει ιδιαίτερα την επιρροή των ευρωβουλευτών. Ε, σίγουρα βέβαια πρέπει να γίνει περαιτέρω μελέτη από του θύματο, γιατί οι μελέτε αυτέ είναι παλιέ. Χρειάζεται σίγουρα επικαιροποίηση. Ο ακαδημαϊκός κλάδο θεωρεί ότι η συμμετοχή αυξάνεται και αυτό συνέβη γιατί υπάρχει ανοιχτό ψηφοδέλτιο, αλλά και γιατί οι ψηφοφόροι μπορούν να κατανοήσουν ότι μέσω του ανοιχτού ψηφοδελτίου μπορούν πραγματικά να αλλάξουν ε, τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ, Γιολάινεν. Äh, vielen Dank. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναλύσεις αυτές. Ήμουν εισηγητής του κανονισμού 2003 του 2003. Μπορώ να σας πω πολλά. Να σας πω ποιες δυσκολίες είχαμε. Και μετά το 2007 εισηγητής για τα ιδρύματα που μπήκαν στον κανονισμό. Χαίρομαι λοιπόν για αυτά τα οποία βρήκατε και διαπιστώσατε. Υπάρχει μια διαφορά της κατάστασης σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. για την εξέλιξη πολιτικών οικογενειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2003 η πολιτική μου οικογένεια ας πούμε δεν μπορούσε να αγοράσει το ένα στυλό γιατί δεν είχε νομική προσωπικότητα ε, ήταν απλά ένα όνομα δεν μπορούσε να πληρώσει το προσωπικό ούτε τίποτα και η πρόοδος με τον πρώτο κανονισμό ήταν πως όλα τα κόμματα τώρα έχουν νομική προσωπικότητα Επίσης θεωρώ πως η έκθεση για να ακούει ήταν μεγάλη πρόοδος. Γιατί δεν έχει νόημα να ε, λέμε πως τα κόμματα μπορούν απλά να εγγράφονται ως ΜΚΟ με βάση το βελγικό δίκαιο. Ε, δεν είναι Greenpeace το κόμμα, είναι μέρος του πολιτικού συστήματος και του δημοσίου χώρου, το είπατε κι εσείς. το μεγάλο ερώτημα που είπατε είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα κατέβουν στις ευρωεκλογές, στον προεκλογικό αγώνα και σε εθνικές εκλογές, σε, σε δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά θέματα σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Το εάν κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο ή όχι. Επίσης το θέμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης πέραν από τον προπολογισμό της Ένωσης. Το 2003-2004 ο φόβος ήταν πως ο Μπερλουσκόνη ή κάποιος άλλος ε, δημοσιο... ε, δισεκατομμυριούχος ή ολιγάρχης ή οτιδήποτε άλλο θα αγόραζε όποιο κόμμα ήθελε. Οπότε είχαμε βάλει ένα όριο ανά άτομο ανά έτος για να μην αγοράζονται κόμματα. Αν δει κανεί πόσα μιμιέ αγοράζονται όμως στα κρατη είναι πραγματικά τρομακτικό πόσα αγοράζουν ε, οι πλούσιοι και τα έντυπα και τα ραδιοφωνικά και οι τηλεοράσεις ανοίγουν σε ένα-δύο άτομα. Ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και ε, θα ήταν ακόμη πιο προβληματικό με τα κόμματα. Το ερώτημα με τα ιδρύματα. Πρέπει να το δούμε. Ρωτήσατε ποιο ενέχει τα ιδρύματα των κομμάτων. μπορούμε να το θέσουμε και εμείς και το και τίθε το ζήτημα και στην ΑΦΚΟ και στο Κοινοβούλιο. Το σκεπτικό ήταν πως τα Ιδρύματα θα γίνουν μια ανεξάρτητη πλατφόρμα ευρωπαϊκού διαλόγου και διαμόρφωσης ε, μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και σύντομα διαπιστώσαμε πως υπάρχουν διαφορές. Ε, κάποια Ιδρύματα είναι πιο κοντά στα κόμματα και στελεχωμένα με κομματικούς ανθρώπους και κάποια άλλα είναι πιο ουδέτερα. Πιο κοντά στα, κοντά στα κόμματα, αλλά ανεξάρτητα. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Επίσης, αυτά τα οποία βρήκατε, δεν ξέρω αν είναι αποστολή των Ιδρυμάτων να συντάσσουν εκλογικά μανιφέστα. Αυτό είναι δουλειά των κομμάτων. και να εκπαιδεύουν για τον προεκλογικό αγώνα. Εγώ το Ίδρυμα το, το θεωρώ ως μια πλατφόρμα διαλόγου, συνείδησης ε, και όχι να αναλαμβάνει αποστολές ε, και τη δουλειά των κομμάτων. Γιατί παίρνουν και τα κόμματα λεφτά από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οι συστάσεις που κάνατε είναι ενδιαφέρουσες. Το εάν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ε, Ευρωπαϊκή, στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Πράγματι αυτό ισχύει όπως και τα συνδικάτα Βεβαίως πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των ακτιβιστών και αυτών οι οποίοι απευθύνονται ε, σε αυτούς. Νομίζω μια αυτοσυγκράτηση λοιπόν των κομμάτων επιβάλλεται. Γιατί μπορεί να υπάρξει και κατάχρηση της ε, πρωτοβουλίας πολιτών και ότι δεν πετυχαίνει κανείς μέσω των εκλογών να προσπαθεί να το φέρει μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. να εμφανίζονται τώρα τα σήματα ναι, στο εκλογικό υλικό, στα ψηφοδέλτια. Ναι, καλό αυτό. Και αυτή η διάκριση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, κάτι ενδιαφέρον πράγματι, αν είναι συμπληρωματική η λειτουργία τους ή αν υπάρχει επικάλυψη. Να μας ενδιαφέρει να μας πείτε πώς έχει αλλάξει αυτό από όταν ε, ξεκίνησε να υπάρχει ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, θετικά αυτά που κάνατε και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτές τις μελέτες. Ευχαριστώ. Ρίτσαρντ Κόρμπετ. Και εγώ ευχαριστώ. Με ενδιέφερε πολύ η μελέτη για τη συνέπεια της τάσης των πολιτικών κομμάτων όχι μόνο ως προς τις ψηφοφορίες αλλά στη στάση τους γενικότερα και τη διαχωρισμό που κάνατε μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Αλλά πώς ακριβώς το ορίζετε, την Ιρλανδία τη βάζατε στο Νότο και τη Μάτα όχι, τη Μάλτα όχι με αυτά τα κριτήρια. Ήταν τρόπος του Λέγιν. θεωρήσαμε ότι η χρήση α, διαφορετικής ορολογίας θα πρόσβαλε μερικούς. Πάλι χωρίς μικρόφωνο ο άλλος τώρα. Τα συζητήσαμε πολύ και τελικά θεωρήσαμε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ουδέτερη ορολογία όπως βορράς και νότος. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ο νότιος, το νότιο τμήμα του κόσμου ή ο αναπτυσσόμενος κόσμος ή οτιδήποτε τέτοιο. Ίσως δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή όπως το δείξατε κι εσείς αλλά αυτή ήταν η λογική μας. ε, τότε τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Γιατί ο ορισμός σας ήταν σωστός. Θα μπορούσε να είχε υπάρξει εκεί πολιτικό, πολιτική διαφορά ή χάσμα. Δεν το περιμέναμε. Α, γι' αυτό είναι ενδιαφέρον. Και συνδέεται, συμβαδίζει με την έρευνα του καθηγητή Simon Hex στο London School of Economics και το συμπέρασμά του είναι ότι οι υποομάδες γίνονται όλο, έχουν όλο και μεγαλύτερη, όχι λιγότερη συνοχή. Αφού όμως αναλύεται κόμματα και όχι απλώς ομάδες στο Κοινοβούλιο, θα έπρεπε ίσως να συμπληρωθούν όλα αυτά και με μια ανάλυση όλων τους των δραστηριοτήτων τα κυριότερα πολιτικά κόμματα οργανώνουν και συναντήσεις προκαταβολικές με υπουργού πριν από τα συμβούλια των κομμάτων τους ή με τους αρμόδιους ή τους δικούς τους επιτρόπους με εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών πολλές δραστηριότητες οι οποίες συνεχώς αυξάνονται πέρα από αυτά που βλέπουμε τόσο ορατά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα. τα κόμματα δηλαδή, όχι στο κοινοβουλίο αλλά γενικά τα κόμματα και το σύστημα του Spitzenkandidaten είναι μέθοδος που, για την οποία πολλοί είχαν αντιρρήσεις αλλά οδήγησε τελικά στην επιλογή του Προέδρου της Κομισιόν. Αυτό νομίζω είναι σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια μελέτη της εξέλιξης των δραστηριότητα των κομμάτων. Ρωτήσατε αν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ εθνικών ιδρυμάτων, think tanks και ευρωιδρυμάτων. Αυτό το ξέρω από τη χώρα μου. Και τα εθνικά επομένως ιδρύματα τελικά καταλήγουν να σκέφτονται λίγο πιο ευρωπαϊκά και αυτό νομίζω είναι επίσης ενδιαφέρον. Αναρωτιέμαι αν τα μικρά ιδρύματα είναι σοβαρά. Αλλά ίσως αυτό να είναι και προβοκάτσια. Τέλος για την πρωτοβουλία των πολιτών δεν νομίζω ότι τα κόμματα θα τη χρησιμοποιήσουν γιατί αν κάτι ένα κόμμα το θεωρεί καλή ιδέα ως κόμμα έχουμε ευρωβουλευτές, έχουμε επιτρόπους δεν χρειάζεται να μαζεύουμε υπογραφές πολιτών και να τις απευθύνουμε στα ίδια όργανα στα οποία έχουμε δικούς μας μέσα. εκτός αν κάνουμε public relations. Ευχαριστούμε Χέλμουτ Σόλτ. Ευχαριστώ. Για να είμαι σύντομος και ακριβής, εγώ δεν είχα την τύχη του Γιολάινεν να είμαι εδώ επί πρώτου ψηφίσματος αλλά συμμετείχα στην έκθεση Γιαννάκου ως και συγητής της ομάδας μας. Και θα έλεγα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση Γιαννάκου θα είχε επιτύχει περισσότερα εάν από την αρχή ήξερε τι θέλει από την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της δομής ε, και της δομής των πολιτικών κομμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση γιατί ε, ανοίγουν εδώ πέρα κάποιες προοπτικές για να συζητήσουμε για το μέλλον και το τι μπορούμε να κάνουμε και δεν έχουμε φτάσει εκεί που χρειαζόμαστε ακόμα. Τέσσερις παρατηρήσεις τώρα. Παραπονιόμαστε όλοι. Το πρωί μιλήσαμε για τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το, τον εκλογικό νόμο πώς θα ε, μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους πολίτες περισσότερο ένα πρόβλημα νομίζω είναι η σχέση μεταξύ εθνικών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών γιατί είναι ένα ζήτημα εξουσίας και κανένα εθνικό πολιτικό κόμμα όσο δεν αναμορφώνουμε το εκλογικό σύστημα, δεν θα συμφωνήσει να δώσει περισσότερη επιρροή, ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οπότε, θα πρέπει να δούμε πώς αυτά θα είναι συνεπή με αυτά τα οποία θέλουν τα ευρωπαϊκά κόμματα ε, και αν δεν γίνει αυτό δεν θα επιτύχουμε. Επόμενη παρατηρήση, συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να είναι τα κόμματα κοινοφελής ε, ενώσεις ε, του βελγικού δικαίου. Πρέπει να υπάρχει μια θεσμική δομή. Έτσι, για να έχουμε και κάποια εξουσία απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Εάν τα κόμματα τώρα έχουν μια δομή ιδρύματος ε, ή θεσμικού οργάνου όπως ε, η Επιτροπή των Περιφερειών Νομίζω θα προχωρήσαμε λίγο παραπέρα. Μετά, η χρηματοδότηση. Από την οπτική των ε, μεγαλύτερων κομμάτων φαίνονται λογικά αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής κερδίσει. Και προς τα εκεί πάνε και οι προτάσεις σας. Αλλά ε, η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα, που είναι διαφορετικό από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ξέρετε πως έχουν πολιτικά κόμματα που δεν έχουν ευρωβουλευτές, πώς ε, μπορούν αυτοί να ε, λάβουν μέρος στη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές προοπτικές κτλ. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και από πλευρά χρηματοδότησης και στην αριστερά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, εμείς δεν είμαστε το κόμμα που θα λάβουμε πολύ ιδιωτική χρηματοδότηση. από μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί, αλλά είναι προφανές. Αλλά ε, ε, δεν πληρώνει εμάς η Gazprom, έτσι εσάς πληρώνει. Λοιπόν... Ε, έτσι και κάπου αλλού που είναι οι πρόεδροι, κάποια άλλη λέσχη που είναι οι πρόεδροι μέλη Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια α, τη λειτουργία ευρωπαϊκών κομμάτων, αν είναι αναγνωρισμένα κτλ. κτλ. Γιατί έτσι υπάρχει και ο ανταγωνισμός για συμμετοχή στη συζήτηση για την περαιτέρω εξέρεξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για τα ιδρύματα Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Άλλη μια παρατήρηση ή πρόταση. Κοιτάξτε, ένα ίδρυμα θα πρέπει να είναι think tank, να εκπαιδεύει, να οργανώνει συγκεντρώσεις ε, για να οργανώνει πολιτικές συζητήσεις, όχι να είναι υποκατάστατο κόμματος αλλά να δίνει στους πολίτες στην Ευρωπαίους να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην δημοκρατική διαδικασία. και έτσι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τον δρόμο και για τις ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες πολιτών. Βεβαίως, ε, οι ευρωβουλευτές είμαστε μεταξύ του πολίτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα think tank νομίζω θα εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης μας. Ευχαριστώ, Μερσέντες Μπρέσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, διότι συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Μια πρώτη παρατήρηση. Επειδή πολλοί από εμά έχουμε ζήσει απευθείας την ε, ποιότητα σε θεσμικό επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, κατά την άποψή μου, παρά τις αδυναμίες τους, έχουν αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να ε, έχουν μια διάρκεια και μέσω των αναλύσεων που μας κάνατε, μέσω των συνηθισμένων κοινοβουλευτικών εργασιών, διότι το να υπάρχει συνένεση μεταξύ ε, ε, ευρωβουλευτών 28 χωρών είναι δύσκολο, αλλά απέδειξαν ότι τα καταφέρνουν και απέδειξαν επίσης και σε αυτή την εκλογική υπόθεση ότι μπορούν να επιβάλλουν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ ε, στενή μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ευρωβουλευτών. Κατάφεραν λοιπόν να επιβάλλουν την απόφαση για τον Spitzenkandidat, κάτι το οποίο δεν ήταν προφανές και επειδή την έχω ζήσει, τουλάχιστον μέσα του Ιδρύματος ε, των Προοδευτικών Σπουδών, έχουν επηρεάσει με το έργο τους, όχι την τελευταία στιγμή, αλλά με ένα έργο ετών, τη δυνατότητα να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Προφανώς η δομή της εξουσίας, τα εθνικά πολιτικά κόμματα είναι πολύ πιο ισχυρά, αλλά ακριβώς ε, διότι υπάρχει μια τάση να αφήνει ανοιχτός ένας χώρος, διότι οι λίγοι είναι ενδιαφερόμενοι για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έχουν καταφέρει όχι μόνο να νομιμοποιήσουν, αλλά να αφήσουν και το χώρο απόφασης και πολιτικού συντονισμού στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία παρά τις αδυναμίες τους κατάφεραν να δημιουργήσουν, τουλάχιστον τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, μία κοινή αίσθηση η οποία είναι προφανής όχι μόνο στα αποτελέσματα, αλλά είναι προφανής και σε όλη την περίπλοκη διαχείριση των συμφωνιών αυτή τη φορά για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, για τις ακροάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να ε, παραμείνει η προσοχή μας στο σημείο αυτό και από αυτό το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί για τον εκλογικό νόμο, προκύπτει ότι η δυνατότητα να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος ευρωπαϊκής κλίμακας, ο οποίος θα είναι αντιπροσωπευτικός των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων, των ευρωπαίων πολιτών και όχι του κάθε κράτος και μέσω αυτών ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και με την ποιότητα ε, της πολιτικής τους επιρροής, τη δυνατότητα πραγματικά να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ των πολιτών των διαφόρων χωρών μελών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, να σκεφτούμε πολύ αυτές τις πτυχές, οι οποίες δεν ξέρω ποιος από εσά, ίσως εσείς ε, κύριε αναφέρατε. Δηλαδή, πέραν των όσων γίνονται εδώ στις Βρυξέλλες, ε, για τους ευρωβουλευτές και για τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Εγώ ήμουν μάρτυρας μιας συζήτησης για την ε, δημιουργία του προγράμματος των σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και οι αρχικές μας θέσεις είχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις και η σύγκληση ε, προς ε, ε, ένα κοινό σύνολο κοινών ιδεών δεν είναι κοινοτοπία, είναι κάτι το οποίο έγινε εδώ με δουλειά στις Βρυξέλλες. Και αυτό συχνά το οποίο μεταφέρεται και σε επίπεδο χωρών, όπου πολύ συχνά τα πολιτικά κόμματα τα οποία κυριαρχούν, τα εθνικά πολιτικά κόμματα, ξεχνούν τι έχουν κάνει και τι έχουν αποφασίσει από κοινού στην Ευρώπη ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το αρνούνται. Επομένως, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και εθνικών πολιτικών κομμάτων, θα πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά προκειμένου να δούμε ε, πως η ε, μετάδοση δεν γίνεται μόνο σε οριζόντιο επίπεδο, αλλά γίνεται και από κάτω προς τα πάνω, αλλά και από πάνω προς τα κάτω. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν λειτουργήσαν και πολύ άσχημα, λαμβάνοντας υπόψη και πόσο ευάλωτα είναι. Σε εμά υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή τη σχέση με τους πολίτες, ήταν η γέννηση μιας ομάδας ακτιβιστών, Ευρωπαίων ακτιβιστών, η οποία προσπαθεί να συμπληρώσει αυτό το κενό. Δεν ξέρω αν συνέβη κάτι αντίστοιχο στα άλλα πολιτικά κόμματα, ίσως θα είχε ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, αλλά έχουμε νέους ενθουσιώδεις υπέρ ε, της ναι, ναι. Ευρώπης που κατάφεραν να ε, δημιουργήσουν ένα δίκτυο ανθρώπων που είναι συνδεδεμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δραστηριοποιούνται στη χώρα τους. Είναι ακόμα λίγοι, αλλά είναι μια καινοτομία που προέκυψε από αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, μία σύντομη ερώτηση. Ήθελα να ξέρω, όταν εξετάσατε όλα αυτά τα ζητήματα, μήπως διαπιστώσατε ότι ε, έχει ενδιαφέρον ακόμα και η ιδεολογία, ε, η εξέταση της νοτροπίας βορράς-νότος κλπ. Ε, αλλά η ιδεολογία προκύπτει σαφώς ως διαφορά στα όλα όσα μελετήσατε. Ο κύριος Μπάντι έχει προκύψει και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων βεβαίως και η μελέτη για τη συνοχή που κάναμε δεν μας δίνει ε, κάποιες μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι θετικό και θεωρούμε ότι κάτι ε, το οποίο είναι πλέον ευρεωμένο ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τόσα χρόνια. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ αναφέρθηκε σε μελέτες οι οποίες έγιναν από τον ε, ε, Higgs στη διάρκεια των ετών και εμείς θεωρούμε ότι τα ερευνητικά δεδομένα για τους ευρωβουλευτές είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικά, διότι... δεν αναφέρει, για παράδειγμα, ότι οι ευρωβουλευτές έχουν μεγάλη πειθαρχία στο κόμμα, κυρίως όταν υπάρχει ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει στις μελέτες μας. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι είναι θετικό ε, το πώς έχει η υγεία των πολιτικών κομμάτων εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Υπάρχουν βέβαια δύο άλλες πτυχές που έχουν εξίσου σημασία. Καταρχάς ε, τα πολιτικά κόμματα έχουν και εξωτερικούς βραχίονες, είναι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πλέον έχουν ε, ένα επίσημο καθεστώς, αλλά επίσης υπάρχουν και τα εθνικά κόμματα και ε, τα εθνικά κόμματα πολύ συχνά είναι ανταγωνιστές. Ε, νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το λέω εδώ αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα της ιδεολογίας ε, έρχεται ε, ε, πιο πίσω, διότι η εθνική ιδεολογία είναι πιο σημαντική. Ναι, ευχαριστώ κύριος Καλόζη. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας για την παρουσία ευρωπαϊκών κομμάτων σε άλλα θεσμικά όργανα. Συνήθως όταν ε, μελετούμε ευρωπαϊκά κόμματα τα χωρίζουμε σε δύο διαφορετικές πτυχές. Υπάρχουν τα θεσμικά και τα εξωκοινοβουλευτικά. Όταν αναφερόμαστε στα θεσμικά έχετε δίκιο. Ίσως επικεντρωθήκαμε υπερβολικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και το πιο σημαντικό θεσμικό όργανο στο οποίο υπάρχει εκπροσώπηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά υπάρχει και εκπροσώπηση και σε, άλλους, ε, σε άλλα θεσμικά όργανα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ίσως θα μπορούσαμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για μελέτη στο μέλλον. Επίσης, ο ρόλος της εσωτερικής δημοκρατίας κάποιο την ανέφερε ή μάλλον κάποιο ανέφερε τη σημασία της ε, ε, υποψηφιότητας του speech and candidate από τα ευρωπαϊκά κόμματα. Ε, και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο επελέγει ο speech and candidate από τα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα. Πέντε κόμμα επέλεξαν υποψήφιο μέσω διαφορετικών κανόνων και η κυρία Μπρέσο προηγουμένως είπε ότι υπάρχει και μια ε, ε, ομάδα νέων ακτιβιστών που δημιουργήθηκε. Ε, κάποιες χώρες χρησιμοποίησαν τις εθνικές τους εκλογές για να επιλέξουν τον... Κάποια, συγγνώμη, πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν τις εθνικές εκλογές για να επιλέξουν τον speech and candidate. Επίσης, Καταλαβαίνω πολύ καλά τις επικρίσεις του κυρίου Κόρμπετ για την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Πολιτών, αλλά ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία είναι ισχυρά και στα θεσμικά όργανα, όπως για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως δεν θα πρέπει να θεωρούν την πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως κάτι το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Όμως θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για να βοηθήσουν τους πολίτες. Από μεθοδολογική σκοπιά τώρα, ναι, δεν είναι η επίσημη ε, απέτηση από το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Ίδρυμα η σύνταξη του εκλογικού μανιφέστου. Εμείς είμαστε πολιτικοί επιστήμονες και ως πολιτικοί επιστήμονες θέλουμε να αναλύσουμε τι ακριβώς συνέβη ε, και πέρα από τον νόμο. Και αυτό ρωτήσαμε στην ερευνά μας ε, στα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά ιδρύματα και στους παλίλους των ιδρυμάτων. Ρωτήσαμε διαδραματίσατε κάποιο ρόλο στην ε, κατάρτιση του μανιφέστου για τις επόμενες ευρωεκλογέ των ευρωπαϊκών κομμάτων και μας απάντησαν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν έχει σχέση με τον κανονισμό, αλλά θέλαμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και όπως είπε και η Μυρσέδες Μπρέσο προηγουμένως, ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων ήταν χρήσιμος πολύ πριν την ε, επίσημη προεκλογική εκστρατεία για να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ των εθνικών κομμάτων που μας έδιναν ε, και αυτά οι ιδέες για τα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, επομένως δύο λόγια να πω. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια για αυτά τα πολύ σημαντικά ε, θέματα, τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των ε, πολιτικών ιδρυμάτων, δεν θέλαμε να δώσουμε την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ε, ε, ψηφίζουν το μανιφέστο και είναι τόσο κοντά στη διαδικασία, γιατί αυτό ε, έχει να κάνει με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αλλά επειδή παρέχουν μακροπρόθεσμη ε, βοήθεια, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν κάποιες ιδέες για το μανιφέστο και να τα χρησιμοποιήσουν και ως εμπειρογνωμοσύνη ερευνητική σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Αντί να ζητήσουν περαιτέρω συμβουλέ, μπορεί να έρθουν να κάνουν κάτι ad hoc. Από αυτή την άποψη λοιπόν θέλαμε να το δούμε αυτό, αλλά ε, η παρατήρησή μα και μάλιστα στη μελέτη, στη ερωτηματολόγιο που δώσαμε στα Ιδρύματα ήταν αν θέλουν να μένουν στην άκρη και να πούνε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα πολιτικά κόμματα είπαν κάποια Ιδρύματα που είπαν όχι εμεί είμαστε κάτι εκ διαμέτρου διαφορετικό και είμαστε απόλυτα διαχωρισμένοι. Θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν τι είναι αυτό και όπω σα είπα η προσδοκία μας ήταν ότι τα μικρότερα Ιδρύματα θα είναι πιο κοντά στα πολιτικά κόμματα και όχι το αντίστροφο διότι αν μικροί ε, ενωθούν, τότε μπορεί να γίνουν πολύ πιο σημαντικοί και να έχουν περισσότερου πόρου στη διάθεσή του. Αλλά τελικώ διαπιστώσαμε ότι ήταν το αντίθετο. Όσον αφορά τη δική σα την ερώτηση, κύριε Κόρμπετ, αν κάνουν κάποια πράγματα τα πολιτικά ιδρύματα και δεν είναι απλώ ε, ε, κα, ε, ε, Έχουμε κάποια στοιχεία στην έκθεση που σας στείλαμε και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα τα κονδύλια, διότι υπάρχουν κάποια ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν για παράδειγμα 200.000 ευρώ ε, προπολογισμό και κάνουν πάρα πολλά πράγματα και κάποια άλλα που είναι σχετικά δρανή ή ε, ε, δεν κάνουν όσα θα έπρεπε. Δεν είναι πάντα θέμα χρημάτων, αλλά θέμα νοοτροπίας και πολιτικών επιλογών. Σας ευχαριστώ. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους που έκατσαν όλους όσοι έμειναν εδώ μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Είναι και η τελευταία συνεδρίαση για τη χρονιά αυτή. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν. Και καλή χρονιά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τους ε, προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρα τις συνεδρίασεις θα τα ξαναπούμε στις 20 Ιανουαρίου όλη η μέρα συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ.